Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αμέσως. Με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν επιφυλάξεις, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρακτικά. Τις προηγούμενες συνεδρίασεις, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, έως το τέλος της συνεδρίασης, θεωρείται πως εγκρινώνται τα πρακτικά. Τώρα θα πρέπει να κάνω κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση. Καταρχάς τα σημεία 10 και 5 της σημερινής διάταξης αντεστράφησαν στη σειρά. Θα αντέστρεψε η γραμματεία λόγω κάποιων ανηλυμένων υποχρεώσεων των ομιλητών μας. Και έτσι το σημερινό υπαριθμόν 5 αφορά την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κένεθ Ντίν. επικεφαλής της μονάδας πολιτικού σχεδιασμού της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ενώ στο σημείο 10 θα γίνει η παρουσίαση του απολογισμού από τον κύριο Ποπόφσκι αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα πρακτικά, για τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης του Συμβουλίου. Και τώρα μπορώ να ξεκινήσω με τις εργασίες μας και το σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Θέμα το οποίο θα συζητηθεί την παρουσία και συναδελφών τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε μικρή συνεδρίαση, καλωσορίζω μαζί τον κύριο Πλέμκοβιτ που είναι εδώ παρόν ω πρόεδρο τη Επιτροπή των Εξωτερικών. Ήθιστε άλλωστε να έχουμε τέτοιε επαφέ και ενημέρωση. Με χαρά καλωσορίζω την εξοχοτάτη Ναταλή Σαπανάτζε πρέσβη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον, την συνοδεύει ο κύριος Ηρακλής Λάτζε. Εκπρόσωπο αμυντικών θεμάτων στην πρεσβεία της Γεωργίας των Βρυξελών. Έχει διατελέσει μάλιστα αρχηγός Γενικού Επιτελείου της Γεωργίας και είχε μια σειρά αρμοδιοτήτων ως στρατιωτικός ακόλουθος στην Ουκρανία, τη Μολδοβία, τη Λευκορωσία, γνωρίζω εκ μέρους της Γεωργίας. Και θα θέλαμε να γίνει η ανταλλαγή απόψεων. γύρω από την πρόσφατη υπογραφή της λεγόμενης συνθήκης στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και αποσχιστικής δημοκρατίας της Απχασίας, από το, από τα εδάφη της Γεωργίας. Και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Σαμπονάτζε να κάνει τις εγωγικές παρατηρήσεις. Και ίσως και ο κύριος Λελάτσα στη συνέχεια. Με συγχωρείτε όμως κυρία μου, θα πρέπει να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πλανκόβιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ποτίκα. Εκ μέρους του Γερμανού Πρόεδρου της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων κυρίου Μπροκ, με χαρά καλωσορίζω την ε, πρέσβη Σαββατνάτζε. Συζητήσαμε άλλωστε και πρόσφατα θέματα σχέσεων της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα το ζήτημα της Νότιας Ουσιατίας και της Απχασίας. Η Επιτροπή των Εξωτερικών φρονεί ότι η υπογραφή της συνθήκης για μια, συμμαχία, ε, για στρατηγική συμμαχία ή με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Αποτελεί μια ανατροπή του status quo. Έχει αντιδράσει τόσο η δική μας πλευρά όσο και το ΝΑΤΟ και θα θέλαμε να ακούσουμε πιο λεπτομερώς από την ε, πρέσβυρα όσο και από τον στρατιωτικό ακόλουθο εδώ στις Βρυξέλλες την αξιολογή τους καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την ασφάλεια της γεωργίας αυτή η συμφωνία αλλά και γενικότερα για την ε, ε, πολιτική γειτονία, την πολιτική την ε, ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να ακούσουμε αν έχετε κάποιες ανησυχίες εκ μέρους της γεωργίας προβληματισμούς αλλά και σχόλια ενδεχομένως για τις εκλογές στη Μολδαβία και την υπερδινιστερία. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία, μάλλον το ζήτημα αυτό της ε, συμφωνίας, στρατηγικής συμφωνίας της ΚΑΚ με την ε, Απχαζία ξεπερνάει τα στενά όρια της περιοχής και φτάνει μέχρι ε, πολύ ευρύτερα επίπεδα που μπορεί να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση, σε, ανα, σε αναζωογόνηση παγωμένων συγκρούσεων και, σε και προβλήματα στην περιοχή. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για την ευκαιρία και να ευχαριστώ σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, για την ε, τεχνητή διοργάνωση αυτής της συζήτησης. Δύσκολη καιρή για τη χώρα μου και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διατεράσσεται η κατάσταση μετά τον ψυχρό πόλεμο, δεδομένου ότι αγνοούνται σύνορα, δικαιολογούνται εισβολές και οι διεθνείς οργανισμοί φαίνονται αδύναμοι. Αυτά ξεκίνησαν με την Απχαζία και την Νότια και την κατοχή τους. Πολλοί πίστευαν εκείνη την εποχή ότι εκεί θα τελείωναν τα πράγματα. Υπήρχε ιστορικό συγκρούσεων στην περιοχή, πολλοί έπεσαν στη σχετική παγίδα, αυτά είναι όλοι κλπ. Αυτό έρεγε ο κόσμος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ό,τι συνέβη στην Γεωργία το 2008 αλλά και προηγουμένως, είναι μια επανάληψη παλαιών γεγονότων. Δυστυχώ είναι κλασική συμπεριφορά μιας συγκεκριμένη χώρας. Η συμπεριφορά αυτή προσβάλλει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασιζόταν η κατάσταση μετά τον ψυχροπόλεμο. Ο βασικός στόχος της παρουσίασης μου σήμερα είναι να σας παρουσιάσω τι τελευταίε κινήσει τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να υπογράψει δηλαδή τη γνωστή Συμφωνία Συμμαχία και Στρατηγική Εταιρική σχέση με τι δύο περιοχέ. Θέλω να εστιαστώ όμω, όχι τόσο στην συνθήκη, τη συγκεκριμένη συνθήκη, η οποία δεν έχει νομική υπόσταση βάσει του Διεθνού δικαίου, αλλά τι ε, διαστάσει που έχει από κοινωνική, νομική και ανθρωπιστική υπόψεω. Επίση να τονίσουμε το πλαίσιο στο οποίο όλα αυτά σοβούν και την ανάλυση των επιπτώσεων για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι γνωρίζετε ότι η συμφωνία, μάλλον μία συμφωνία, η οποία τίθεται σε ισχύ σε συνδίκε στρατιωτική κατοχή δεν έχει κανένα νόημα και αντίκρισμα. Αυτό συμβαίνει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι προθέσει της Μόσχας είναι απολύτω σαφεί αν κάποιο είχε αμφιβολίες. Λίγα λόγια για το περιεχόμενο τη συμφωνία, τη συνθήκη, μάλλον. Πρόκειται για, για συντονισμό πολιτική, πολιτική πολιτικής ασφάλειας και άμυνα συμφωνίε για αμοιβαία προστασία σε περίπτωση εισβολή. Κοινό έλεγχο των συνόρων, κοινέ περιπολίες στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ενίσχυση των συνόρων με τη Γεωργία και άνοιγμα συνόρων με τη Μητροσική Ομοσπονδία δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου με την προσάρτηση της Απχαζίας στο κοινό σύστημα ασφαλείας της νότιας περιοχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εισαγωγή του ρωσικού κανονιστικού πλαισίου μεταξύ άλλων και τελωνιακών δασμών. Προοπτική ενσωμάτωση της Επικραζίας στο ρωσικό σύστημα. Δημιουργία κοινών πολιτιστικών και ανθρωπιστικών ε, δεσμών Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο αυτό που θα περιλαμβάνει και εναρμόνιση της ε, εκπαιδείας. Λέει επίση η συμφωνία ότι όλες οι οικονομικές πτυχές της ε, υλοποίησης αυτής της συμφωνίας θα καλυφθούν από την Ρωσική Ομοσπονδία. Όλοι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα πληρώνονται από την Ρωσία βάσει του Μισθολογίου της Νότιας Ομοσπονδίας περιοχή της ε, Ρωσίας. Αυτό ισχύει και για τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνησή μου χαρακτήρισε αυτήν την συνθήκη ως βήμα προς την προσάρτηση της ε, Χαζίας και αποτελεί μια περαιτέρω προσβολή της εδαφικής ανεξαρτησίας και κυριοτητας της, της Γεωργίας. Θέλω ευχαριστήσω και για άλλη μια φορά την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μου δίνει. Υπάρχει λοιπόν το διεθνέ δίκαιο, αλλά υπάρχουν και άλλε συγκεκριμένε επιπτώσει στην περιοχή. Η συνθήκη δημιουργεί αυτό το οποίο η Ρωσία ονομάζει νέα πραγματικότητα στο πεδίο. Όπω έγινε με την ε, Κρυμαία, με, την, το διαχωρισμό εδαφών, ε, πράγματα τα οποία είναι τελεσμένα γεγονότα και είναι δύσκολο να ανατραπούν. Αυτό κάνει και η συνθήκη με την Απχαζία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Απχαζία ουσιαστικά εγκαταλείπει την ε, ούτως ανεξαρτησία της ανεξαρτήτως του θέματος της νομιμότητας ή όχι που είχε δημιουργείται επίσης ένα ισχυρότερο σύνορο με την γεωργία δεν ξέρω αυτό αν θα είναι τείχος ή απλό σηματοπλέγμα το συνολικό μήκος των σηματοπλεγμάτων στα σύνορα είναι 50 περίπου χιλιόμετρα, περίπου 50 χιλιόμετρα. Διαιρείται έτσι και η γεωργική υγεία αλλά και ο πληθυσμό τη περιοχή. Κάποιοι, μάλιστα τον τοπικό πληθυσμό, εγκαταλείπουν αναγκαστικά τα σπίτια του. Στην Αφγαζία, από τον Ιούνιο του 2013 οι δυνάμεις κατοχής ξεκίνησαν να σκάβουν ορίγματα, να δημιουργούν ε, οχυρωματικά έργα ενισχύοντας την οχυρωματική συνορική γραμμή. Τα ορίγματα αυτά είναι 3 μέτρα βαθιά και έχουν πλάτος 4 με 5 μέτρα. Επίσης, ε, σημαίνει δηλώνει τα σύνορα στο μέσο της γεωργικής γης. Η συμφωνία αναφέρεται σε περαιτέρω ενίσχυση αυτών των συνόρων, το οποίο σημαίνει ότι εντός δύο ετών από την θέση σε ίσχυ μπορεί πραγματικά να προκύψει μια πραγματική, ένας πραγματικός διαχωρισμός της επεργασίας από την υπόλοιπη γεωργία. Αυτό σημαίνει ενισχυμένου ελέγχους στην διακίνηση του πληθυσμού, περισσότερα σημεία ελέγχου, παρενοχλήσεις ε, και απαγορεύση των τοπικών πληθυσμών. Αυτό οδηγεί, με οδηγεί στο δεύτερο σχολείο μου για τις ανθρωπιστικές δηλαδή επιπτώσεις της συμφωνίας. Δεδομένου ότι με τα κινήσει του πληθυσμού γίνονται όλο και πιο δύσκολε. η πρόσβαση σε υγεία και άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε στη Γεωργία ε, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη για του κατοικού τη Απχαζία. Όσοι φέρουν διαβατηρία, οι γεωργίε θα έχουν περισσότερε δυσκολίε στην Απγαζία. Επίσης, θεμελιώδη δικαιώματα όπω η γλώσσα και η παιδεία ε, θα είναι λιγότερο προσιτά. Η συμφωνία δεν κάνει καμία αναφορά στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ακόμα και η γλώσσα της Απχαζίας αναφέρεται περιστασιακά και μόνο εν παρόδο στην συμφωνία. Η συμφωνία επίσης μειώνει τις πιθανότητες να βρεθεί διαπραγματευ... λύση μέσω διαπραγματεύσεων και επίσης υπονομεύει κάθε πιθανότητα για τη Γεωργία να έχει απευθεία διάλογο με την Απχαζία. Η κυβέρνηση της Γεωργίας υιοθετεί μια ανοιχτή πολιτική και έχει προσπαθήσει να συνομιλήσει απευθείας με τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος ε, αποκόπηκε με βίαιες μεθόδους από την υπόλοιπη Γεωργία. Μετά από τη συμφωνία, η πολιτική συμμετοχή και διαπραγμάτευση που είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Με ποιους θα μιλήσουμε, με ποιους θα διαπραγματευτούμε και με ποιο σκοπό και με τι αποτέλεσμα. Μας ενισχύει επίσης πολύ μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις στις ομιλίες της Γενέβης που είναι ο βασικός μηχανισμός για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ειρήνευσης και Κατάπτωσης του Πυρός του 2008. Φοβούμε μάλιστα ότι η συμφωνία αυτή θα παραλυφθεί και θα αφορά και άλλες χώρες της περιοχής εκ των πραγμάτων προσάρτηση της περιοχής θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην διαδικασία στην περιοχή. Η συμφωνία είναι απειλή όχι μόνο για την ανεξαρτησία και δαφική κυριότητα της Γεωργίας αλλά και για την ασφάλεια της περιοχής και της Ευρώπης γενικότερα. Βλέπουμε μια εκθετική αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στη Ρωσία στην περιοχή. Η Ρωσία χρησιμοποιεί μάλιστα τις στρατιωτικές της δυνάμεις με τρόπο βρυδικό μη ορθόδοξα έλεγα, κάτι οποίο αποτελεί περαιτέρω απειλή για την ασφαλεία. Η προσάρτηση της Κρυμαίας και τώρα της Απχαζίας στην πράξη δείχνει την στάση της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα. Για τη Γεωργία αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανασφάλεια καθώς το στρατιωτικό προσωπικό εξοπλισμός και πυρομαχικά συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στα σύνορά της. Θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα στρατεύματα της Ρωσίας που σταθμεύουν στην περιοχή για τις στρατιωτικές βάσεις και το καθεξής αλλά αυτό θα το κάνω αν χρειαστεί και ίσως απαντώντας ερωτήσεις στην Αμπχαζία και στην ευρύτερη περιοχή οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις είναι τουλάχιστον τρεις η Ρωσική Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή συνεχίζει να εξοπλίζει αυτές τις βάσεις όλο και περισσότερο με νέα άρματα μάχης και επιθετικά οπλικά συστήματα Ενισχύοντα, όπω είπα, τι δυνάμεις κατοχής. Πέρα από τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων, η Ρωσία ανακαινίζει και αναπτύσσει νέε μεταφορικέ υποδομέ στην περιοχή, κατά το οποίο θα τις επιτρέψει να μετακινεί τι δυνάμεις τη ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τέλο, η κατάσταση που περιγράφω έχει επιπτώσει που εκτείνονται πέραν της Απχαζίας και της περιοχής. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση διεθνών αρχών και κανόνων, κάνουν την κατάσταση λιγότερο προβλέψιμη και αυτό καταστρέφει την βάση για όλες τις ε, ειρηνικές διαπραγματεύσεις που έχουμε τώρα στην περιοχή. Οι αρχές για τις οποίες μιλάμε δεν είναι θεωρητικές αρχές, έχουν σχέση με την ασφάλεια στην περιοχή. Η πρόθεση του διεθνούς δικαίου προστάτευσε μικρά κράτη από εισβολές στο παρελθόν. Και αυτό γινόταν μέσω τη κοινή επιθυμίας όλων των ε, κρατών, μελών τη διεθνού κοινότητας, να αποφύγουν τέτοιου είδου προηγούμενα. Έτσι, καταφέραμε να συνέσουμε έστω και σιπηρά σε διεθνεί κανόνε. Το παραβίαση των συνόρων και η εδαφική ακυρότητα είναι ένα από αυτού του κανόνε που έχει παραβιαστεί και όχι μόνο μια φορά. Αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο για μας που θυόμεθα αμέσω, αλλά και για το σύστημα γενικότερα. Τα προηγούμενα δυστυχώς επαναλαμβάνονται και μάλιστα με τρόπο μη προβλέψιμο. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν στη Γεωργία το 2008 αποτέλεσαν προηγούμενο για την Ουκρανία και την Κρυμαία το 2014. Το πλαίσιο διαφέρει βεβαίω κάθε φορά, όμω τα αποτελέσματα και οι περαιτέρω επιπτώσεις ε, παρουσιάζουν μεγάλε ομοιότητε. Και στι δύο περιπτώσει, μια τρίτη χώρα χρησιμοποίησε στρατιωτικά μέσα για να καθορίσει τι πολιτικέ επιλογέ μια άλλη κυρίαρχη χώρα. Και στι δύο περιπτώσει, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνδυασμό πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών πιέσεων. Και στι δύο περιπτώσει, η άμεση εμπλοκή τη τρίτη χώρα σαν τη αντίσταση. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν υβριδικά μη ορθοδόξα μέσα και άλλε στρατιωτικέ δυνάμεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα από σταθεροποίηση και πίεση. Η εισβολή στο τέλος υποτίθεται ότι υποστηρίζεται από το επιχείρημα της προστασίας του πληθυσμού και των αρχών που εν τέλει παραβιάζονται κατάφορα. Αυτό συνέβη, επαναλαμβάνω, όχι μία φορά, αλλά δύο. Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι το ερώτημα πλέον στο μυαλό μα είναι ποιανού είναι τώρα η σειρά. Για να επανέλθω στο θέμα τη ε, συνθήκη, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία είπε δεν υπάρχει τίποτα καινοφανέ εδώ και δεν καταλαβαίνουμε, λέει, γιατί όλη αυτή η φασαρία. Η δήλωση αυτή του Υπουργού Εξωτερικών ε, είναι αληθή, αλλά και <laughs> αναληθείς. Δηλαδή είναι ακριβές από τη μια πλευρά ότι τα όσα μόλις περιέγραψα δεν είναι απλώς ένα χαρτί το οποίο υπεγράφει μία εβδομάδα πριν. Είναι αποτελέσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας που ξεκίνησε τον ρόλο της Ρωσίας ως ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή και που κορυφώθηκε το 2008 με την εισβολή της Γεωργίας, στη Γεωργία και κατάληψη της Απχαζίας. Από τότε η Ρωσική Ομοσπονδία κατάφορα γνώρισε την ειρηνευτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την διαμεσολάβηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να αποσύρει τα στρατεύματά τη από τη Γεωργία, αναγνώρισε και τι δύο υποκατοχή περιοχέ ω ανεξάρτητα κράτη. Έτσι φτάσαμε στην Συμφωνία Φιλίας και Αμοιβαία Αρρωγή. Το 2009 ακολουθήθηκε αυτό από άλλα κείμενα που ενίσχυσαν τον έλεγχο της Απχαζίας. Το 2010 οι στρατιωτικές βάσεις της ε, Ρωσίας επέξαν επίσημη υπόσταση. Επίσης δεν είναι κοινοφανές ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται φυσικά για την ανεξαρτησία τη μια ή τη άλλη περιοχή. Ποτέ δεν ήταν ένα έντιμο διαμεσολαβητή στην περιοχή. Αυτό το οποίο όμω είναι κοινοφανέ εν τέλει είναι ότι τα προσωπία πλέον πέφτουν και γίνονται σαφεί οι προθέσει τη Ρωσία. της τη αλλη περιοχη ποτε δεν ηταν ενα εντιμο διαμεσολαβητη στην περιοχη αυτο το οποιο ομω ειναι κοινοφανές εν τελει ειναι οτι τα προσωπια πλεον πεφτουν και γινονται σαφει οι προθεσει τη ρωσια η ρωσια καταπατησε την ανεξαρτησια τη απχαζιας στο κέντρο εισαγωγικών και δεν αποκρύβει πλέον τις προθέσεις της να ενσωματώσει την περιοχή αυτή στον πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ρωσίας. Βασικά η Απχαζία είναι πλέον μέρος της νότιας ομόσπονδης περιοχής της Ρωσίας. Είναι επίσης νέο ότι η κατοχή του αυτό ήταν απάντηση στην πρόταση της Γεωργίας. Η Γεωργία να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό παντά ακριβώ και η πρόσφατη κίνηση το 2008. Η Ρωσία λέγει ότι το ΝΑΤΟ πηλεί την δική της ανεξαρτησία. Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία. Και αυτήν τη θέση ορισμένοι εν μέρει έστω την κατανόησαν. Η Ρωσία την εποχή εκείνη παρόλα αυτά είπε ότι δεν είχε μια αντίρρηση. Τα πράγματα σήμερα όμω άλλαξαν. Οι δράσει τη Ρωσία στην Μολδαβία, την Ουκρανία και τώρα στην Απχαζία και τη Γεωργία δείχνουν ότι η Ρωσία έχει τελικά αντίρρηση για οποιαδήποτε ακίνηση η οποία δεν είναι υπό τον ελεγχό τη. Σα καλώ να αξιολογήσετε τώρα και με τη σειρά σα την κατάσταση στην περιοχή και να υπερασπιστείτε τι αρχέ των οποίων υπεραμείνεται πάντα η Ευρώπη. στο επικείμενο ψήφισμα για την ε, Γεωργία. Παρακαλώ να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αναλάτσο θα λάβει το λόγο για να απαντήσουμε μετά και σε ερωτήσεις. Και ξε... Α, όχι, δεν θα λάβετε το λόγο, οπότε ξεκινάει η συζήτηση. Παρακαλώ τους συναδέλφους να περιορίσουν τις ε, τοποθετήσεις τους στα δύο λεπτά. Ο κύριος Καρίν πρώτα. Αντιπροσωπεία για τη σχέση με τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη σαφέστατη παρουσίαση της κατάστασης όπως ε, διαγράφεται. Ασφαλώς και προσυπογράφω όλα όσα υπόθηκαν ιδιαίτερα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Προοπτικής και της δικής μου όταν λέτε ότι πρέπει να ε, σταθεί η Ευρώπη αντιμέτωπη με όποιον χρειάζεται για να στηρίξει τις αξίες τις οποίες προασπίζεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τη Γεωργία αλλά και γενικότερα θα ήθελα να διερευνήσω κάτι στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς ε, εν συντομία στην τοποθέτησή σας. Ένα κείμενο που κυκλοφόρησε σε σχέση με τη λεγόμενη Sbedlim Society θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους και βλέπουμε κάποια διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο ρωσικό κείμενο. Είχα χτες μια συνεδρίαση με τον πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο Σάλβα, που είχα οργανώσει εγώ. Θα ήθελα λοιπόν για όλους εμάς εδώ να δούμε τη δική σας εκδοχή των πραγμάτων, διότι τα κείμενα είναι διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία και κατά τρόπο πολύ σημαντικό. Διαβάζοντας τα λοιπόν, μπορεί κανείς να καταλήξει το συμπέρασμα ότι κάποια στοιχεία της ε, κοινωνίας της Απχαζίας τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα από αυτή που παρουσιάζει η Ρωσία. Τα στοιχεία αυτά πώς τα βλέπει η Γεωργία και τι θα συμβούλευε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επαφές της, στις σχέσεις της με τα στοιχεία αυτά. Ο κύριος Πλάνκοβιτς παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Φορτίγκα. Και εγώ ήθελα να κάνω αντίστοιχη παρατήρηση και ερώτηση με τον κύριο Καρίμ, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δύο εκδοχές του κινημένου. Θα χρειαζόταν περισσότερη σαφήνεια, λοιπόν, για να δούμε ποιο είναι ουσιαστικά το επικρατούν και σε τι συμπεράσματα πρέπει να καταλήξουμε. Και επίση, για να συμπληρώσω τόσο από τις ομιλία σα, θεωρείτε ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί μια απόπειρα για ε, de facto οριστικοποίηση, επισημοποίηση της προσάρτησης Απχαζίας από την Ρωσία. Ευχαριστώ, Στέτινα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για τη Γεωργία τώρα τελευταία. μετά από όριμη σκέψη και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της σύνταξης αυτού του κειμένου ήταν η Νότια Σετιακή και η αστικά έχουν καταληφθεί αφού μετά από προσπάθεια απόσχησης και εμείς προσπαθήσαμε με τους συναδέλφους ώστε το ψήφισμα αυτό να μην περιέχει την έκφραση περιοχές που επιθυμούν να αποσχιστούν. Έτσι. Και νομίζω ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ καλό είναι να λέμε τα πράγματα εδώ με το πραγματικό του όνομα Κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε τον σωστό ορισμό και ε, στην Αμχαζία το, την αρχή της δεκαετίας του 90 και αυτός ο τότε πρόεδρος της που ήταν υπέρ της απόσχησης ε, συνεργαζόταν με μία ομάδα Ρώσων ε, εκεί επί τόπου και υπήρχαν ένοπλες ρωσικές ομάδες με στρατιώτες ε, με μπλεμπερέ ε, που έφερναν όπλα στους ε, ντόπιου προσπαθούσαν να αποσχεστούν Εδώ έλεγαν ότι εδώ κανονικά ήταν μια κατάληψη κλασικής μορφής μιας περιοχής χώρας άλλης, διαφορετικής. Και εδώ δεν ξέρω, αλλά αν ε, δεν ε, κάνουμε κάτι όλα αυτά που ξεκίνησαν με την Απχαζία, με την Τσετσενία, μετά με την Νότια Ασετία με την Κρυμαία, βλέπουμε τη σειρά αυτή. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και στα ανατολικά της Ουκρανίας και όλα αυτά θα μπορούσαν ακόμη περισσότερο να συνεχιστούν. Άρα λοιπόν να λέμε το όνομα, με το όνομά τους τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να παρακαλέσουμε εδώ να κρατήσει την υπόσχεσή του και να δούμε ποιες είναι ακριβώς οι βάσεις και να ξέρουμε και οι στρατιωτικές δυνάμεις που είναι στην Απχαζία, πόσες είναι. Ναι, δίκιο, δίκιο έχετε σχετικά με αυτόν τον όρο που, το, που κανονικά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε. Μαρκόρα. Ναι, σας, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους από τη Γεωργία για την ενημέρωση και να πω ότι η Απχαζία είναι ένα βαρόμετρο για την περιοχή. Βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σύραξης που οφείλεται στη Ρωσία. Ακόμα και οι διάφορε αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις, στις υπηρεσίες ελέγχονται από τους Ρώσους. Δεν θυμάστε και του Ολυμπιακού στο Σότσι. Μετά μετακινήθηκαν τα σύνορα για να δοκιμάσουμε τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Το μόνο το οποίο έγινε ήταν η ενίσχυση των δυναμένων κατοχής. Σήμερα η Ρωσία βλέπει τη Δύση και τον ΝΑΤΟ ως εχθρό εναντί του οποίου υιοθετεί επιθετική συμπεριφορά. Εμείς ως πότε θα βλέπουμε τη Ρωσία ως εταίρο. είναι του οποίου υιοθετούμε φιλική στάση. Θα προστατεύσουμε τους ε, πραγματικούς εταίρους μας από τις επιθετικές βλέψεις της Ρωσίας. Πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε εδώ τους φίλους από την ε, Γεωργία και ε, δυσκολεύομαι να ομολογήσω αυτό, αλλά η αντιδράση μας στην αρχή της κρίσης ήταν ανεπαρκής. Το ομολόγω αυτό. Και έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Χθες συζητήσαμε την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί λιγότερο αν θέλετε παθητική. Εάν δεν εξεύρουμε πιστική λύση για να αντιμετωπίσουμε τη συμπεριφορά της Ρωσίας, είναι βέβαιο ότι θα γίνουμε μάρτυρες περαιτέρω επιθετική συμπεριφοράς, εισβολών, εις βάρος ακριβώς των φίλων μας. Αλλά και εμείς θα βρεθούμε σε όλο και πιο δύσκολη κατάσταση. Συνεπώ. αντί για περισσότερα λόγια, κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι στην πράξη. Να επιταχύνουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, τις, τη δράση μας. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, έχω ένα μακρύ καταλογό ομιλητών. Πρέπει να κλείσει ο καταλόγος των ομιλητών, ο κ. Σαν Ήθελα να σας ευχαριστήσω Τρέφουμε συμπάθεια στη Γεωργία για την κατάσταση αυτή. Δυστυχώς όμως όλα αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Και ο πρέσβης της Ρωσίας έχει δίκιο. Η Ρωσία έχει καταλάβει τα τμήματα αυτά και δεν θα τα εγκαταλείψει εύκολα. Και η Ρωσική Ομοσπονδία βέβαια προσπαθεί να προσαρτήσει τα εδάφια αυτά. Και και για τους επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, τι θα γίνει ε, τι μπορούν να μας συμβολεύσουν, τι μπορούμε να κάνουμε για να σταθεροποιηθεί τουλάχιστον η κατάσταση και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί η κυριαρχία σας εκεί. Ευχαριστούμε κύριε Λαζού. Ε, με συγχωρείτε δεν κατάλαβα την προφορά του ονόματός μου. Λοιπόν, ε, μάλιστα, η κατάσταση είναι σαφής, ε, την επιβεώνει η πλευρά της Γεωργίας. Εγώ έχω προκαταβολικά ενημερωθεί βεβαίως, ε, έχω διαβάσει και παλαιότερες εκθέσεις και την έκθεση της Επιτροπής του 2009 όπου είναι κάπως διαφοροποιημένη η εικόνα που παρουσιάζεται. Γιατί φαίνεται από την έκθεση αυτή ότι είχε διαπράξει το πρώτο βήμα προς τον πόλεμο, προς την πολεμική αντιπαράθεση Γεωργία. Την ερμηνεία αυτού του θέματος δεν θέλω τώρα να την αναλύσουμε, αλλά ερωτώ πώς πάμε από εδώ και μπρο. Υπάρχουν προσπάθειες αυτές οι χαμένες περιοχές, οι αποσχιστικές περιοχές όπως θέλετε να τις ονομάζετε, να ανακτηθούν. Γιατί νομίζω πως είναι γεγονός ότι μετά τον πόλεμο οι περιοχές αυτές έχουν προσανατολιστεί ακόμη πιο έντονα προς τη Ρωσία. Δεν αρκεί η ερμηνεία η Ρωσία έχει κατοχή πάνω στις περιοχές αυτές. Ερωτώ λοιπόν, από εδώ και μπρος τι γίνεται. Γίνεται διάλογος για το να εξασφαλιστεί για τις περιοχές αυτές εγγύηση μη επίθεσης μακροπρόθεσμα ή ε, εξακολουθεί να ε, υπάρχει ο κίνδυνος της απόπειρα να ανακτηθούν με στρατιωτικά μέσα οι περιοχές αυτές. Υπάρχουν κάποιες εγγύσει. Ευχαριστώ. Κύριος Μπουστινάρου. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Την κυρία Πρέσβη θα ήθελα να την ευχαριστήσω για όσα μας είπε. Είναι πραγματικά δραματικές αυτές οι εξελίξεις. Δεν είναι όμως κάτι το καινούριο. Είναι βέβαια μια καινούρια φάση της όλης ρωσικής στρατηγικής. Την έχουν ενορχιστρώσει υπέροχα και μετά βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν στρατιωτικά μέσα για να έχουν ένα πλήρη έλεγχο σε μια περιοχή που όσον αφορά το διεθνές δίκαιο είναι κατηλημένη περιοχή. Εντάξει, όποιο όρο θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και επίση από στρατηγικής πλευράς. Πρόκειται βέβαια για ένα νέο μονοπάτι που ακολουθεί η Ρωσία και σίγουρα θα εφαρμοστεί και αλλού αυτό. Ε, εντάξει. Εδώ θα πρέπει να τα δούμε αυτά πραγματικά σοβαρά και να καταλάβουμε ότι και στην Ουκρανία την Ανατολική και εκεί θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η νέα στρατηγική. Πρόκειται για μια επιθετική στρατηγική. Πρόκειται για μια δράση επιθετική και που αποσταθεροποιεί την περιοχή εκεί αλλά και την όλη ισορροπία την περιφερειακή και όχι μόνο τοπικά. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε όσους τρέφουν ακόμα αυταπάτες ότι η Ρωσία η οποία έχει Ρώσους υπηκόους σε άλλα εδάφη μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και να ακολουθήσει και δεύτερη φάση και τρίτη φάση και αυτό αποσταθεροποιεί την περιοχή. Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Για την εξαιτημή κυρία Πρέσβυρα και τους υπόλοιπους θα ήθελα να απευθύνουν ερώτημα. Οι ρωσικές δυνάμεις στην Κρυμαία, πώς βλέπετε τα πράγματα, είναι για να αλλάξει η σχέση εκεί γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα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 αναμφίβολα. Αυτά τα δύο μέρη που καταλαμβάνονται είναι μια ρήξη, αλλά θα πρέπει να δούμε το ρελισμό μας τον πολιτικό, τον υπάρχοντα στην περιοχή εκεί. Ας ρίξουμε μάτια η νομιμότητα ότι θα προσαρμοστεί στην πραγματικότητα όταν η πραγματικότητα έχει τέτοια σημεία εκεί. Ίσως υπάρξει μια ρήξη περί του λογικού της υπόθεσης και εδώ και 50 χρόνια ας πούμε το Ισραήλ ε, προχωράει σε ρήξη της διεθνούς νομιμότητος ε, και με τετελεσμένα γεγονότα και υπάρχει μια διαφορά όμως ότι στο Ισραήλ κανείς δεν το κυνηγάει, εν τη Ρωσία ναι. Εδώ 50 χρόνια συμβαίνουν πολλά πράγματα και δεν λέει κανείς τίποτα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι η δύναμη είναι πραγματικότητα, ισχύς επιτόπου και πολλές φορές καλύπτεται αυτή η πραγματικότητα, αγνοείται. Υπάρχει μια βασική διαφορά για μένα ανάμεσα στη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Εσείς ε, τι έχετε, μια εθνική πραγματικότητα σταθερή συμπαγή υπέρ του αραγούς αυτού του εδαφικού και σχετικά με άλλες εκλογές στην Μολδαβία και στην Ουκρανία. Εδώ τι έχει γίνει από τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ρωσία για την αναγνώριση της εδαφικής ακυρότητας ε, και της Ουκρανίας ε, και παντού γύρω όλων των εδαφών αυτών έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή από πλευρά Ρωσίας ε, που σιγά σιγά προχωράει σε αυτά τα εδάφη. Τι ακριβώς γίνεται και αυτή η ρωσική αντίληψη για να προχωρήσει τα πολιτικά και στρατιωτικά σύνορα και για τη Γεωργία που θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ και εκεί που το θεωρούν σαν, εθνικό, σαν έδαφος ασφαλείας. Ε, ας πούμε έχουμε στον Παναμά που βλέπουμε την ε, εισβολή εκεί όταν υπήρχε απειλή. Κύριος Φραντζολίτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ουδέν των νεότερων από το Ανατολικό Μέτωπο. Γιατί δεν ξεκίνησε το 2008. Το 1991-1992 ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Όταν ξέσπασε η πρώτη σύγκρουση. Θερμή πρώτα, μετά με μετατράπησε ψυχρή όπως και οι λοιπές και ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο με συγκρούσεις που μεταμορφώνονται σε ψυχρές, καταψύχονται, αλλά μπορεί και να αποψυχούν και να φτάσουν μέχρι σημείο βρασμού ανά πάσα στιγμή. Πρόκειται για ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, για περιοχές που βρίσκονται γύρω από τη Ρωσία και φαίνεται δυστυχώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στη να αντιμετωπίσει επαρκώς τις απειλές και προκλήσεις της Ρωσίας. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασία με τον ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί ότι μια συνολική στάση και πολιτική απέναντι στην πολιτική της, ε, την επιθετική πολιτική της Ρωσίας είναι απαραίτητη. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ήδη να αναπτύσσεται αυτέ τι μέρε. Πρέπει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και τον ΝΑΤΟ να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται να πάψει αυτή η επιθετικότητα τη Ρωσία και δεν μπορούμε τη ρωσική πολιτική να την αντιμετωπίζουμε μόνο με δηλώσει, μόνο με λόγια. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, ξέρετε. Έχουμε να κάνουμε με μια νέα υβριδική μορφή ψυχρού πολέμου εν εξέλιξη. Πρέπει να επιβάλλουμε νέε κυρώσει. Πρέπει να λάβουμε νέα στρατιωτικά μέσα και να αντιδράσουμε. Και όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα που θα αντιμετωπίσουν αυτά που συνεχίζει να κάνει στην Ευρώπη η Ρωσία. Πριν δώσω τον λόγο και πάλι στην κυρία Πρέσβη, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ασφάλεια του ξύλου θα προσταθεί στη ημερησία διάταξη και θα συζητηθεί μαζί με το θέμα της ασφάλειας στην Βαλτική. Θα έχουμε δηλαδή ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα από διαφορετική βεβαίως οπτική γωνία, ευρύτερη πάντως. Οπότε από την πλευρά μου προς το παρόν σύμφωνο με πολλούς από τους προλαλήσαντες ότι δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική μορφή πολεμικής σύραξης η οποία όμως ήταν ήδη ορατή εδώ και χρόνια. Ήρθε όμως σήμερα η ώρα να κάνουμε κάτι για να την αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πρέσβη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα σχόλια και ερωτήσεις που ακούστηκα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο εξαντλητικά. Θα αναφερθώ καταρχάς στη διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων και τις αντιδράσεις από την κοινωνία, την αφχαζική κοινωνία για τη λεγόμενη αυτή συνθήκη. Πολύ σωστά υπήρξε μια προηγούμενη, μια πρώτη συνθήκη όπου μιλούσε μάλιστα για ολοκλήρωση, για ενοποίηση. Τώρα μιλάνε για συμμαχία και στρατηγική εταιρική σχέση. Η πρώτη αυτή εκδοχή του κειμένου ήταν που οδήγησε σε έκφραση δυσφορίας συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου της του λεγόμενου Κοινοβουλίου της Απχαζίας που συζήτησε με βάση μια προφορική ερώτηση το θέμα. Πολλοί Απχαζοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, θεώρησαν ότι πάει πολύ μακριά ότι είναι υπερβολική αυτή η συμφωνία και θέλησαν να εισαγάγουν κάποιες αλλαγέ. Όντω εισήχθησαν κάποιες αλλαγέ. Πιστεύω όμως ότι είναι μόνο εξουραϊστικού, τύπου. Δεν υπάρχει πέραν της αλλαγής στον τίτλο καμία διαφορά σε σχέση με το τελικό κείμενο το οποίο έχω εγώ μαζί μου και μπορώ να σας δώσω γιατί ουσιαστικά στο κείμενο μέσα γίνεται λόγος για ενοποίηση της, η ένταξη της ε, Απχαζίας στην κοινωνικό πολιτική και στρατιωτική σφαίρα επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης γίνεται λόγος ε, για την ε, διευκόλυνση ως προς την χορήγηση της λεγόμενης ηθαγένειας, της απχαζικής ηθαγένειας σε Ρώσους πολίτες, δεν ξέρω αυτό στην πράξη, αλλά πάντως υπήρξαν και γι' αυτό αντιδράσεις. Είδαμε κάποιες αλλαγές λοιπόν για να ολοκληρώσω, αλλά το τελικό κείμενο που έχω εγώ, η τελική έκδοση που έχω στα χέρια μου, ουσιαστικά μιλάει για, αποτελεί μάλλον μία συνθήκη de facto προσάρτησης. Γιατί ακόμη και αν είχε αναγνωρίσει ε, την ε, ψευδοανεξαρτησία η Ρωσία της Απχαζίας τώρα ουσιαστικά προχωράει σε προσάρτηση κάτι το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί εάν προχωρήσει Πολλοί από σας ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα πρέπει να εμπλακούμε, ποια είναι η συνταγή. Εγώ και ταξινομικές συνταγές δεν έχω να σας δώσω, είναι πολύ περιπλοκή η κατάσταση. Το βήμα όμως αυτό, έστω και αν δεν είναι πρωτόγνωρο, γεννά νέα δεδομένα και εισάγει νέες διαστάσεις σε μια κατάσταση ήδη δύσκολη. Και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ανατραπεί, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στην φάση πριν από την εμπλοκή. Αυτό που κάνει η Ρωσία ουσιαστικά είναι να καθίσταται εγγυητής της μη διευθέτησης της σύγκρουσης. Για πολλά, χρόνια δεν είχαμε πραγματικές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία με την απχαζική πλευρά. Χωρίς πολιτική και στρατιωτική επέμβαση από τρίτο κράτος. Το τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι μόνο θεωρητική ε, ερώτηση. Δεν ξέρουμε τι έχει συμφωνηθεί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει από τη συμφωνία αυτή, ε, αλλά πάντως δεν διευκολύνει τη λύση. Και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί εμπλέκεται και παρεμβαίνει η Ρωσική Ομοσπονδία με αυτόν τον τρόπο. Η πρόοδος βέβαια στη συνθήκη υπερπλέκει ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Είπαμε ήδη ότι οι κυβερνητικές δομές Απχαζίας μπαίνουν υπό την αιγίδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ε, το, το σύνολο της δίκης του στρατού, τα, ο έλεγχος των σύνορων, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με πραγματική ε, υλική, υλικό διαχωρισμό της Απχαζίας από τη Γεωργία. Ναι, μπορεί να, είναι, να μην είναι κάτι το καινούριο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε σε αυτό, γιατί είναι όλη αυτή η λογική ακριβώς που μας εμποδίζει. Όλοι λένε, α, παλιά ιστορία, το ξέραμε, ας το προσπεράσουμε. Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι με την αποδοχή ενός τετελεσμένου εμφανίζονται νέες πραγματικότητες, οι οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς θέλησα να έρθω να σας μιλήσω. Γιατί μπορεί να μην είναι πρωτόγνωρη αυτή η ιστορία, αλλά είναι ένα επιπλέον βήμα, σημαντικό βήμα που δεν πρέπει να λησμονούμε. Και πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι η χώρα η οποία πραγματοποιεί τα βήματα αυτά τα πραγματοποιεί ενώ την παρακολουθεί απραγεί η διεθνή κοινότητα γιατί δεν έχει στη τη διεθνή κοινότητα σημαντικά εργαλεία όντω δεν είναι εύκολο να τοποκριθεί κανεί στι προκλήσει που ε, συνεπάγονται οι δράσει τη Ρωσία αλλά έχουμε καθόλου να αναλογιστούμε τι είδου ε, απαντήσεις ή αντιδράσεις μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να έχουμε έτοιμες απαντήσεις. Γιατί αυτό θα συμβεί πάντοτε είναι η ίδια η εικόνα, ε, ανεξαρτήτως του τι συνέβη ε, το 2008 και ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά δεν θα συμφωνήσω βέβαια με την εκτίμησή σας, γιατί την ε, Γεωργία την προκάλεσαν να μπει στον πόλεμο αυτό και άλλωστε ε, υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Και ναι, βεβαίως πρέπει να ρωτήσουμε και τον απχαζικό πληθυσμό, αλλά η πλειονότηση του απχαζικού πληθυσμού που ζούσε νόμα στην Απχαζία έχει εκτοπιστεί, έχει απελαθεί και άρα έχουμε να κάνουμε με μια, με μια γενετική εκαθάριση, μια φυλετική εκαθάριση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πρέπει, εάν είναι να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, να είναι σε θέση να επιστρέψουν στι ε, αιστείε του και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων. Ιδάλω η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ άδικη. για τις πραγματικότητες, ε, για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην ε, περιοχή, το, την ε, Ρωσία και την προσπάθεια για την εξασφάλιση μιας ζώνης επιρροής που παραβιάζεται κατά τη θεώρηση την Ρωσική από το ΝΑΤΟ. Ναι, δεν πρέπει να λησμονούμε τους υπολογισμούς της Realpolitik που μπορεί να ε, προκάλεσαν ακόμη οι ανατροπές αυτές, τις οποίες έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως έχουμε να κάνουμε με 25 χρόνια από την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του ψυχρού πολέμου και όμως υπάρχουν κράτη τα οποία ακόμη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι γίνονται ανεκτά κάποια κράτη, θα πρέπει να γίνονται όλες οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανεκτές των αντίων. Θα πρέπει να καταδικάζονται πάντοτε. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από ένα κράτος θα πρέπει να οδηγεί πάντοτε, δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί άλοθη για την μη καταδίκη άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Και επίσης ζούμε σε μια διαφορετική αντίληψη. Η αντίληψη που έχει η Ρωσία για τη ζώνη επιρροής της είναι μια αντίληψη πολύ παλαιωμένη του ψυχρού πολέμου για να μην πω του 19ου αιώνα. Απαρχαιωμένη. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αυτήν ως μια ρυθμιστική δύναμη, θα πρέπει αυτή την ρύθμιση ή την ε, επιβολή ε, των ε, κανόνων των αρχών να ε, ψώνει το ανάστημα και να την υπερασπίζεται όταν παραβιάζονται οι κανόνες και οι αρχές. Και εδώ δεν μιλάμε για επέκταση του ΝΑΤΟ. Η Γεωργία όντως προσπάθησε να καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν τα κατάφερε. Εδώ μιλούμε για προσέγγιση και μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για επιλογές. Επιλογές του λαού μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι χώρα θέλει να είναι η Γεωργία και σε ποια χώρα θέλουν οι Γεωργιανοί να ζουν. Το ότι βρισκόμαστε κατά τύχην στην λάθος σφαίρα επιρροής δεν μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε κατά κάποιον τρόπο που εμείς δεν επιλέγουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. κύριος Τζινιλάντζε θέλει και αυτός να συμβάλλει. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ δύο λόγια για τις ε, κινήσεις της Ρωσίας σε σχέση με τη Γεωργία και τα στρατεύματα που έχει αναπτύξει. Έχουμε περίπου 4.200 Ρώσους, 200 στρατιώτες στη μία περιοχή και 4.500 στην Απχαζία. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης 1.325 στο Σλοβάλι συνοριοφύλακες και άλλους 1.325 συνοριοφύλακες στην Απχασία Το σύνολο 11.250 περίπου Ρώσοι στρατιώτες. εγκαταστημένοι στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας στην περιοχή Σκυβάλη με την τέταρτη λεγόμενη στρατιωτική βάση της Ρωσίας βλέπουμε εξοπλισμό νέο, σύγχρονο προηγμένο 15 τεθαρακισμένα, 160 οχήματα του πυροβολικού, 900 APC, μεγάλους όλμους, συστοιχίες πυροβολικού, και προηγμένο εξοπλισμό, Αντιαεροπορικά όπως τα ΠΟΚ, τα Τότσικα, ελικόπτερα Ατόκε, ΕΜΑ24. Στην Απχαζία δε έχουμε επίσης 50 τεθωρακισμένα T90 νέας φουρνιάς, 125 μαχητικά οχήματα, 160 επίση τέσσερις μεραρχίες Χάουιτσερ αντιεροπορικά συστήματα και πυράβλους S300. Και μια μεραρχία βαλιστικών πυράβλων καθώς και μαχητικά ελικόπτερα Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ρωσία διατηρεί μεγάλο αριθμό δυνάμεων και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού στα κατεχόμενα εδάφη ικανό να στηρίξει στρατιωτική επιθετική δράση κατά της γεωργίας. έχει περιθώριο δε 48-72 ώρων για την ενίσχυση των στρατευμάτων αυτών από το Βόρειο Κάφκασο. Μία πολιτική μόνο απόφαση του Κρεμλίνου θα αρκούσε για την οργάνωση προκλήσεων από την άλλη πλευρά της κατοχής, της ρωσικής κατοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ακόμη ένα πρόσχημα για πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσινολάτσε. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο, πολύ σύντομο, γιατί έχω και εγώ μια ερώτηση προς την ε, κυρία Πρέσβη. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι ε, η κατάσταση και πώς έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες της Γενέβης. Θα θέλαμε τις δικές σας θέσεις. Και επίσης, Οσετία και Απχαζία εσωτερικός εκτοπισθέντες. Ποια είναι η κατάσταση σχέση με αυτούς. Ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη μέρημνα για το θέμα αυτό η Γεωργία και καθώς έχω και εγώ προσωπική πείρα, οι άνθρωποι αυτοί ξέρω ότι η πατρίδα τους θεωρούν την Απχαζία και την Οσετία. Αντίστοιχο. Και εκεί θέλουν να ζουν όσο καλή αντιμετώπιση και να έχουν στη Γεωργία. Στόχος τους είναι η επάνωδο στις αιστείες τους. Δεν αναπτύσσουν μία μόνιμη εγκατάσταση εκεί που βρίσκονται. Είναι προφανές αυτό και τώρα θα παρακαλέσω αν θέλει κανείς να συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των συζητήσεων. Mr. Castaldo, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την αξιότιμη κυρία Πρέσβη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα λεπτομεριακά που μας είπε μια εκτίμησή της ε, για όλη αυτή την εικόνα. Μου φαίνεται ότι αλλάζουν ε, εντελώς τα πράγματα στη Μαύρη Θάλασσα και Πούτιν το Κρεμλίνο. Ε, το South Stream δεν θα το πραγματοποιήσει πια. Και από την Κωνσταντινούπολη ένα καινούριο αγωγό μάλλον προς την Τουρκία μετά προς το Αζερμπαϊτζάν βλέπουμε ότι υπάρχουν εντάσεις με την Αρμενία επειδή πριν από μερικές εβδομάδες βλέπουμε ότι κατερριφθεί ένα ελικόπτερο και επίσης τρίτο στοιχείο στην Ολυσκακέρα Έχουμε αυτή τη γοητευτική, ας την πούμε έτσι, συμφωνία με την Αμχαζία, μια ρήξη στον Κάφκασο. Η δική σας εκτίμηση της εικόνας ποια είναι, υπάρχει κίνδυνος παρέμβαση της Ρωσίας μαζικά. Εκεί ή πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός για να δείξει ότι υπάρχει ένταση σχεδόν λίγο πιο κάτω από την κόκκινη γραμμή αλλά να έχει δύναμη έτσι για διαπραγματεύσεις. Ναι, ο επόμενος και μετά θα κλείσουμε τον κατάλογο. Υποστηρίζοντας τις προτάσεις του συναδελφού Καστάλντο, Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί η ένταση στρατιωτική πρωτό, άμεσα με τη Ρωσία, εκεί, στην Οσετία και δεύτερο, μέσω της Αρμενίας που είναι σημαντικότατη στρατιωτική βάση της Ρωσίας ε, εκ των πραγμάτων. Δύο uwagi. No po pierwsze to mm, bardzo tu niepokojąca jest ta informacja mm, o wojskowym Θέλω να πω ότι αν δούμε το που μπορεί να πάει η Ρωσία, τι μπορεί να κάνει η Ρωσία. θα ανησυχούμε διότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα ακραίας δράση. αλλά αυτό ένα άλλο ερώτημα. Αντιθέτως, τι δυνατότητες έχουν οι ένοπλες δυνάμεις της Γεωργίας. Η Ρωσία γνωρίζουμε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά η Γεωργία ε, δεν ξέρω, έχει ενισχύσει καθόλου τις δυνάμεις της ε, μετά από τη σύραξη με την Ρωσία. Κυρία Πέζες. ευχαριστώ. Όσον αφορά τις συνομιλίες στη Γενέβη, πολύ σημαντικές για μας, γιατί είναι ένα διεθνές σχήμα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε την σύραξη. Δύσκολα τα πράγματα, οι συνομιλίες ε, δεν πηγαίνουν πάντοτε κατευχήν. Συζητήσαμε και την περασμένη φορά εστιάζοντας στα πιο προβληματικά σημεία όπως τη δημιουργία τεχνητών συνόρων και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στον τοπικό πληθυσμό. Κάτι άλλο σημαντικό όσον αφορά τις συνομιλίες στην πρώτη μας εργασία. Η Ρωσία έχει υποσχεθεί να πόσχει από χρήση στρατιωτικής δύναμης και όμως αυτό συνέβη. Η Ιωρία στην Γενέβη αυτό δεσμεύτηκε να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη και περιμένουμε, προσδοκούμε να κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Και όμως αυτό όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά η Ρωσία εντείνει τη στρατηγική παρουσία στην Απχαζία και την Οσιτία. Επίση, στην ομάδα εργασία 2, ανθρωπιστικά ζητήματα. Ανησυχούμε για τι επιπτώσει. Ανέφερα την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα. Συζητήθηκε και αυτό. Ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι επίση ε, η επιστροφή των εκτοπισμένων, των ιστορικά εκτοπισμένων. Οι εκπρόσωποι της Εκπραζίας που ελέγχονται από τη Ρωσία βεβαίω ε, δείχνουν μια προθυμία να συζητήσουν το θέμα. Η κατάσταση των εκτοπισμένων πάντως γενικά στην ε, Γεωργία είναι προβληματική. Έχουν βρεθεί προσωρινά καταλήμματα, αλλά όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για προσωρινή λύση για κάποιους, να μην υπάρχουν αυτές οι λύσεις. Αντιμετωπίζουμε κύματα Πάντω και έχουμε αντιμετωπίσει κύματα εκτοπισμένων τη δεκαετία του 1990 μέχρι και το 2008. Λόγω πάντω τη ύπνωσης αυτού του τεχνητού συνόρου αυτό το σηματόβλεγμα για το οποίο σα μίλησα το αποτέλεσμα σύνορο εντός, αυτό, εισαγωγικών αυτό να περνάει μέσα από τις αυλές σπιτιών ε, κάνοντα τα πράγματα αδύνατα για κάποιους κατοίκους. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει υποστηρίξει στην προσπάθεια αυτή. Είναι βοήθεια για την οποία η κυβέρνηση της Γεωργίας είναι ευγνώμων. Όσον αφορά την παρουσία της Ρωσίας τώρα στον Εύξηνο Πόντο και το τι σημαίνει για την ασφάλεια, την ισορροπία δυνάμεων και το καθεξής. Είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς. Και δεν ξέρουμε ως που θα πάει η χρήση στρατηγική δύναμης από τη Ρωσία. Ένα είναι η Ρωσία κατ' επανάληψη απέδειξε την πρόθεσή της, την πράξη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό έγινε για πρώτη φορά με τρόπο κατάφωνο στην Γεωργία το 2008 και το να υποστηρίζει κανείς ότι δεν θα ξαναγίνει δεν να σου πω νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα το 2008 αλλά και σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας καταφορής εισβολής με χρήση στρατιωτικής δύναμης από τη Ρωσία εις βάρος γειτονικής χώρας. Έγινε μία φορά και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ξαναγίνει. Εξαρτάται ποια θα είναι τα κίνητρα και ποια θα είναι η στόχη της Ρωσίας. Η κατάληψη της Κρυμαίας και τώρα ο έλεγχο επί της Απχαζίας αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων, εννοείται στον εύξηνο πόντο. Το αν αυτό είναι μια προσωπική κίνηση ή δημιουργία νέου status δεν ξέρω. Πάντω η Ρωσία προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι κυρίαρχη δύναμη στον εύξηνο πόντο. και περιμένει, προσδοκά ότι οι κινήσεις αυτές θα γίνουν, ε, θα τύχουν αντίδραση σε πολλές χώρες. Ναι. Εδώ ε, διδασκόμεθα από το 2008 και έχουμε προσαρμόσει τα προγράμματά μας και την αντίληψή μας στρατιωτική για να έχουμε ικανότητες ε, σε μια στην όλη μάχη και να μπορέσουμε να έχουμε και μια αντιροπορική άμυνα, ένα κατάλληλο έλεγχο και η κύρια προσπάθειά μας αφορά μια διαδικασία που θα σημαίνει αλλαγές στις ειδικέ δυνάμεις για δυνατότητες μάχημας επιτόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η της πρέσβης και του στρατητικού εκπροσώπου του στρατητικού συνδέσμου ας μας θα χρησιμοποιηθούν για να αποφασίσουμε να προκρίνουμε μία στάση εδώ και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σίγουρα η αντιπροσωπεία μας θα συνεχίσει τη σχετική συζήτηση. Ε, κύριε Πέτζη, θα είμαστε σε επαφή. Σφαλάντζε, θα είμαστε σε επαφή εννοείται και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Παρακαλώ, παρακαλώ, στις θέσεις σας. Θα μπορούσατε να παραμείνετε στις θέσεις σας, παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Ladies Κυρίες και κύριοι. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Εδώ θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Κένεθ Ντίν, καλώς ορίσατε. συμμετείχε ήδη σε μια συνάντηση της Επιτροπής που είχε σαν θέμα τις πολιτικές αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΕΛΕΞ που με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πολιτικές αποστόλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που είστε εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Έχετε αναλάβει την, την όλη στρατηγική σχετικά με το σχεδιασμό αυτό. Ήρθα να σας μιλήσω για τις ε, τέσσερις ε, αποστολές ε, πολιτικής προστασίας που έχουμε και αυτές που θα αναπτυχθούν στο επόμενο χρόνια θα προσπαθήσω να σας ε, μιλήσω στους δυνατόν ε, πιο συνοπτικά και να ακούσω στη συνέχεια τις ερωτήσεις σας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τις ευρωπαϊκές αποστολές με την τελευταία αυτή που αφορά την Ουκρανία η οποία θεσπίστηκε τον Ιούλιο εφέτος, αλλά ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο, το Δεκέμβριο, πριν από τρεις μέρες, AU, AM, Ουκρανίας, λοιπόν, με τον κύριο Μισέ, επικεφαλής, μια αποστολή που στόχο έχει να προσφέρει να αρρωγή στις Ουκρανικές αρχές και με στρατηγικές σύμβουλες σε σχέση με τα ζητήματα στο Κίεβο. Περιορίζεται ακόμη στο Κίεβο, δεν βγαίνει ακόμη έξω από το Κίεβο. Έχουν συνομιλήσει τα κράτη-μέλη, κατά τρόπο υγιή θα έλεγα, για το σχεδιασμό. Σε ένα χρόνο θα πρέπει να γίνει ανασχεδιασμός και επανεστίαση ενδεχομένως, ανάλογα και με τις θέσεις των κρατών μελών. και την εστίαση ενδεχομένως ε, και έξω από το Κίεβο. Πάντως ο στόχος είναι η χρηστή διακυβέρνηση, η ελαχιστοποίηση της διαφθοράς σε επίπεδο κυβερνητικό, δικαστικό, αστυνομικό, ανθρώπινα δικαιώματα, προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο αστυνομεύεται ο Ουκρανός πολίτης, ευρωπαϊκές πρακτικές, λογοδοσία, δημοκρατική και δημόσια λόγοδοσία προς τον πολίτη. Αρχική διάρκεια της αποστολής είναι δύο χρόνια, με αναθεώρηση όπως είπα πάνω στο χρόνο για να ε, γίνει επανεστιασμός εάν χρειαστεί, 13,8 εκατομμύρια ευρώ με 101 σε διεθνές επίπεδο και 75 σε τοπικό επίπεδο υπαλλήλους. Κοσμοπέδιο. Μια από τις πιο παλιές μας αποστολές. Όπως και πρόεδρος τη Δευτέρα είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτές τις αποστολές ενώπιον της Επιτροπής των ε, Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και του των προϋπολογισμών. Ιδιαίτερα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με αστυνόμευση σε όλο το κοσφοπέδιο, αλλά ιδιαίτερα στο Βόρα. Μια σημαντική ευαίσθητη και πολιτικά περιοχή, αλλά σημαντική ιδιαίτερα και για την ενότητα του κοσμοπεδίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με διαχείριση συνόρων, με τελωνιακές υπηρεσίες, τελωνιακό έλεγχο, εισαγωγή αστυνομικών προδιαγραφών, μια εντολή η οποία επειδή δεν ήταν εξατλητική και αρκετά σαφής ε, οδήγησε σε δυσκολίες στην εκτέλεση, γιατί έπρεπε να αναμειχθούν κάποια στοιχεία υποχρεωτικά με μη δεσμευτικά, αλλά με τελική απόφαση των κρατών μελών τον Ιούνιο του 2016 θα κλείσει πιστεύουμε το θέμα αυτό. Άρα έχουμε τα δύο τελευταία ε, χρόνια. Και άρα έχουμε ακόμα 14-15 μήνες για την αποστολή αυτή. Έχουμε ένα κύριο στοιχείο, την ειδική ομάδα κρούσεως για τις έρευνες, η ITF, που εδρεύει στις Βρυξέλλες μεν, αλλά κυρίως δραστηριοποιείται στο Κωσυφοπαίδιο με εκθέσεις από το 2011 επί παραδείγματι που μιλούν για την ε, λαθροδιακίνηση ανθρώπων ή εγκλήματα πολέμου όπως απαγωγές, φόνοι και διερευνά τέτοια ε, περιστατικά όπως αυτά που συνέβησαν το 1999 στον πόλεμο μπορεί να οδηγήσει σε προσαγωγές στο δικαστήριο στις κάτω χώρες οι οποίες ήδη έχουν ε, αναλάβει να υποδεχθούν. Και έτσι το 2015 θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη δουλειά αυτής της Task Force, η οποία βέβαια έχει ψηλό προϋπολογισμό με 180 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια και με τους περιορισμούς βέβαια στην οικονομία που γνωρίζουμε. Το επόμενο θέμα είναι η EUMM στη Γεωργία που μόλις συζητήσατε, άρα θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία. Πρόκειται για μια αποστολή από το 2008, συμφωνία μεταξύ Μετιέτευ και Σαρκόζη, έξι σημείων που στόχο είχε να γίνει σεβαστό το σύνολο των έξι σημείων της συμφωνίας από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι η αποστολή, 200 παρατηρητές για την Νοτιοσετία και την Απχαζία. Πρόκειται για μια αποστολή που έχει γίνει αποδεκτή, πιστεύω. Πρόκειται για μια απασχολή που εξυπηρετεί καλές υπηρεσίες, ε, ακόμη και την αποτροπή διάδοσης ψευδών ειδήσεων για το τι λέει μια πλευρά εις βαρός άλλη, της άλλης, είναι κάτι το ευπρόσδεκτο πιστεύω τις γεωργιανές ε, αρχές, χωρίς να ξέρω τι υπόθηκε στο προηγούμενο κομμάτι της συνεδρίας σας. Πάντως είναι πολύ σημαντικό μέσον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της σε σχέση με τη γεωργία και την ευρύτερη περιοχή. Ένα μέσον που ονομάζεται Instant Prevention Reporting Mechanism άμεσος μηχανισμός ε, ενημέρωσης IPRM που αναπτύσσεται στην Νότια Οσιτία αλλά όχι ακόμα στην Απχαζία και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει προσπάθεια για αποτροπή της συνεργασίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχών εκεί. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα περάσματα τα συνοριακά. Ε, ορίζουμε προτεραιότητες για την εξομάλυνση, για τα μέτρα εμπιστοσύνης, για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την αποτροπή το, της επανέναρξης των ε, εχθροπραξιών με αποστολή καταρχάς δύο χρόνια και άλλα δύο προσθέθηκαν συνέχεια. Στη Μέση Ανατολή έχουμε τη Γιούπολ Κόπ στη Ραμάλα με 71 μέλη διεθνή προσωπικού ε, διεθνούς προσωπικού, 1,8 εκατομμύρια. Ξεκίνησε το 2006, πρόκειται για μια από τις πιο παλιές αποστολές. Επικεντρώνεται στην ε, Παλαιστινιακή Διοίκηση, στη Δυτική ε, Όχθη. Ουσιαστικά υπάρχει, υπάρχει πρόβλεψη και για την Γάζα, αλλά μόνο στην Δυτική Όχθη μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες της προσπάθεια για αναμόρφωση του δικαστικού, την επιβολή του κράτους δικαίου, συνεργασία με τα δικαστήρια, τους δικαστές, ενημέρωση και κατάρτιση της αστυνομίας. Επτά σχολές αστυνομικές στην ε, πλευρά που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή με σημαντική επιτυχία στην κατάρτιση της Παλαιστινιακής Πολιτοφυλακής. Η Γιούμπαμ Ράφα είναι μια πολύ μικρή αποστολή, βρίσκεται εν υπνό ουσιαστικά. Με 980.000 ευρώ, περιορισμένο προσωπικό, λίγο πολύ λειτουργεί από το Τελαβίβ ε, και περιμένει να επαναδραστηριοποιηθεί με την κατάπαυση, ε, την καταλλαγή περισσότερο στην περιοχή. Ετοιμάζουμε ένα έργο προετοιμασίας όπως το λέμε, προπαρασκευής. Δηλαδή προπαρασκευάζουμε την Παλαιστινιακή Αρχή να ξαναγυρίσει στη Ράφα, στη Γάζα και αυτή είναι η δουλειά μας, ιδιαίτερα όσον αφορά το ε, σημείο διάβασης της Ράφα. Κοιτάμε από ευρωπαϊκής πλευράς να δούμε τι, τι πρέπει ακόμα να γίνει για να υπάρξει ουσιαστικό άνοιγμα του περάσματος της ράφα. Βέβαια ξέρετε ότι οι πρόσφατες αποστολές έκαναν ε, μια απόπειρα να καταγράψουν τι άλλο μπορεί να γίνει ε, για να σημειώσει την παρουσία της η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γάζα γενικότερα ε, και όταν είναι όριμες οι συνθήκες θα μπορέσουμε να απτύξουμε τις ε, δραστηριότητές μας αλλά και θα χρειαστούμε και περισσότερο προσωπικό και περισσότερα στοιχεία ασφαλείας. Και προχωρώ. Στην Αφρική, UCAP Sahel Mali, που θεσπίστηκε το 2014 η δέκατη αποστολή που ξεκινάει 15-16 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται τώρα η προπαρασκευή της στα κεντρικά γραφεία για να δούμε με ποιους θα συνομιλήσουμε, σε ποιο τομέα θα κινηθούμε. Πάνω απ' όλα πάντως θα επικεντρωθούμε στην αναμόρφωση των αστυνομικών αρχών, της εθνοφυλακής, σομαλικής και του Μαλή έχουμε ιδιαίτερα τη μηνύσμα, δηλαδή την ε, δύναμη σταθεροποίησης, συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και στη Νέα Υόρκη αλλά και ε, με τις επιτόπου ε, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών για να μην υπάρξει επικάλυψη και από την 1η Ιανουαρίου θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην διοίκηση, την αστυνομία, τις, ε, τους ανθρώπινους σπόρους, τις προδιαγραφές, την λογοδοσία στον Παμάκο που θα επισκεφθώ όταν είναι δυνατόν για να μεταφέρουμε, ε, βρίσκονται τα γραφεία μας, ε, θα προσπαθήσουμε όμως όταν είναι όριμες οι συνθήκες να τα μεταφέρουμε στα βόρεια, εκεί που είναι πραγματικά η ανάγκη εφόσον βεβαίω ε, το επιτρέψουν οι συνθήκε. Τα κράτη-μέλη τώρα θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε στον Παμακό. Αλλά βέβαια οι συνθήκε ασφαλεία είναι πολύ σημαντικέ και πρέπει να αναπτύξουμε συνεργατικέ δράσει και οικονομία κλίμακα βεβαίω και μια κοινή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ανατολικά πάω τώρα, Ιούκαπ Νέστο, νότια ανατολικά. Έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια στις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Συνεργαζόμαστε με την Άβο Ατλάντα. Νέα στρατιωτική αποστολή, θαλάσσια στρατιωτική αποστολή στον ε, Ινδικό ωκεανό, το κέρας της Αφρικής. Για λόγους ασφαλείας καταρχάς επικεντρωθήκαμε στο Τζιμπουτί με κατάρτιση της λιμενοφυλακής της ακτοφυλακής, ενημέρωση για το τι μπορεί να συμβαίνει στη θάλασσα και εφαρμογές στη στεριά, διάφορες υπηρεσίες ε, που προσφέρονται σε πέντε χώρες, την Σομαλία, την Κένια, το Τζιμπούτι, την ε, Σαϊσιέλ και το Τζιμπουτί επιλογή των κρατών μελών ήταν να επικεντρωθεί η αποστολή στην Σομαλία. Προς το παρόν, για το 2015, ξεκινάμε λοιπόν με ένα μικρό ε, γραφείο με 6-7 συναδέλφους στην Σομαλία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνεργασία και με τις δικαστικές αρχές και μετά, με ένα, και μετά συνεχίζουμε με ένα μικρό γραφείο επίσης στο Μογκαντήσου, 5-6 άτομα που ελπίζουμε να διευρυνθεί αργότερα έτσι ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Συνεργαζόμαστε με τις αντιπροσωπείες και τους ειδικού απεσταρμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θέλουμε να γίνει ως το δυνατόν πιο ε, πλήρης και ολιστική η προσέγγιση. Η Γιούπολ Αφγανιστάν Ιδρύθηκε στις 17 Ιουνίου του 2007, αν δεν απατώμε, με προσωπικό διεθνές. Έχει τώρα μπει στα τελευταία δύο της χρόνια. Έχουμε επανεστιαστεί σε τρεις γραμμές δραστηριότητας για το 2014. Την συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της αστυνομίας του Αφγανιστάν, μεταρρύθμιση του Υπουργείου των Εσωτερικών, και για να είμαι ειλικρινής, είχαμε πολύ σαφή και έντονη παρουσία αμερικανική στο Αφγανικό Υπουργείο των Ιστορικών και χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι καλύτερο το Υπουργείο Ιστορικών να έχει πολιτική διοίκηση και να διοικεί σωστά τις αστυνομικές του δυνάμεις και να συντονίζει την υποστήριξη από το στρατό όπου χρειάζεται να υποστηρίξει τις αστυνομικέ αρχές και βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ε, το πλέγμα σχέσεων της αστυνομίας με τις αγγελικές αρχές. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και το αστυνομικό σύστημα, το σύστημα ανακρίσεων της αστυνομίας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να περάσει συντοχρόνω στις αγγελικές αρχές. Άρα λοιπόν 10 Δεκεμβρίου του 2016 τελειώνει αυτή η, αποστολή, η εντολή αυτής της αποστολής. Τώρα βρισκόμαστε στο Χαρατάν, στο Μαζισρίφ, στη Βόρεια, στη βόρεια χώρα, στο Βόρειο Αφγανιστάν, με γερμανικές δυνάμεις εγκατεστημένες πρόκειται να αποσύρθουν το 2015 και άρα θα παραμείνουμε εν τέλει και για το τελευταίο στάδιο στην Καμπούλ. Εντοπίζουμε επίσης προβλήματα σχέση με την ε, ε, τήρηση του κράτους δικαίου για να εστιαστούμε σε επόμενο στάδιο και θέλουμε να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία δραστηριοτήτων για το στάδιο μετά το 2016. Εν τέλει, η Γιούμπαμ Λιβύης, μια αποστολή δύσκολη, ε, εξ αρχής θεσπίστηκε το Μάιο του 2013, έχει εντολή μέχρι το Μάιο του 2015. Θα είσαστε όμως και εσείς ενημέροι ότι έχει μετατραπεί σε πολύ δύσκολο περιβάλλον αυτό της Λιβύης στις 22 Νοεμβρίου. Αποφάσισε αν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν το προσωπικό μας στα 17 μέλη διεθνούς προσωπικού που για ένα μήνα προσπάθησαν όσο μπορούσαν να εντοπίσουν αξιόπιστους και σοβαρούς ε, συνομιλητές για την αποστολή αυτή που αφορά τη διαχείριση των συνόρων, αλλά δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν γιατί δεν υπήρχαν αξιόπιστοι συνομιλητές. Προσπαθήσαμε και στην Τρίπολη της Λιβύης και στην περιοχή του αεροδρομίου. Η κατάσταση όμως δεν επέτρεψε να προχωρήσουμε όπως θα θέλαμε. Έχουμε γύρω από τη Μίτκα, από τη Μιστράτα, γύρω από το αεροδρόμιο δυνάμεις ε, των Ηνωμένων Εθνών που διατηρούν την τάξη και που μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξή τους. Πάντως, Κάπου στις 16-17 Δεκεμβρίου πρόκειται να εκφραστούν ε, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και ίσως κάποια κράτη-μέλη εκφράσουν πιο, ε, με πιο μεγάλη ακρίβεια τους στόχους τους και τις προθέσεις τους. Εμείς θέλουμε να μείνει η αποστολή στο δυνατόν περισσότερο στην ε, Λιβύη. 26,2 εκατομμύρια ευρώ. Κοστίζει και Πρόεδρε, νομίζω ότι πέρασα πολύ γρήγορα τις αποστολές μας, αλλά αυτές ήταν εν όλο οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διοικητά, και τώρα παίρνουμε σε ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Ντρογιεύσκη, καταρχήν. Το πρώτο ερώτημα είναι δημοσιονομικής φύσης. Είμαστε περί τα τέλη της χρονιάς. Ερωτώ λοιπόν, έχουμε προϋπολογισμό ή τις 9,5 αυτές αποστολές. Στο Μαλί το κόστος αυξάνεται. Στη Λιβύη, στη Λιβύη πετύχαμε να εξοικονομήσουμε κάποια κονδύλια αλλά θα μπορέσουμε να κινηθούμε στα πλαίσιο του προπολισμού του 2014. Και τώρα Ουκρανία Κίεβο είναι μια αποστολή η οποία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται στην ανασκόπηση των εκλογών. Ποια είναι η αποψή σας παρακολουθούμε ικανοποιητικά την κατάσταση συμπεριλαμβανομένου του Ντόνμπα. Και δεν λέω για την κατάσταση στον στρατιωτικό τομέα, λέω για την υποστήριξη προς τον πληθυσμό, προς τους πολίτες. Διότι η κυβέρνηση σταμάτησε κάποια προγράμματα υποστήριξη, εδώ δεν πληρώνει οι συντάξει. Λοιπόν, είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε αποτελεσματικά την κατάσταση. Και κάτι άλλο. Είπατε για ένα μηχανισμό άμεσης αντίδραση στην Γεωργία. Τι εννοείται, τι είναι αυτό ο μηχανισμός. Διότι μόλις ακούσαμε για την ε, στρατιωτική εμπλοκή μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας στη Γεωργία. Έχουμε 10.000 ε, στρατιώτες στην περιοχή, βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό, άρματα μάχης ε, και άλλα οπλικά συστήματα. Μιλούμε για μια επιθετική δυνατότητα μεγάλη κλίμακα. Εμεί με ποιο μηχανισμό θα αντιδράσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο νάρτ. Σνάρτ. Ορισμένες για μερικέ αποστολέ. θα θέλω να υποβάλω. Εκεί από τη στιγμή που το Ισραήλ ε, δεν ε, έχει τον έλεγχο της καταστάσεως ε, εκεί ακριβώς που απαγόρευσαν και την είσοδο από τους φιλελεύθερους ας μιας αποστολής η κυβέρνηση του Ισραήλ που λέει ότι από τις... έχει πολλές και καλές σχέσεις μαζί μας και απαγορεύει στους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού που υποστηρίζουν ε, την Γάζα. Και εκεί την είσοδο επιτόπου την απαγόρευσαν. Γιατί σε ένα παρόμοιο να έχουμε μια αποστολή. Δεύτερο, στο Αφγανιστάν. Λέτε ότι η αστυνομία, η δικαιοσύνη θα πρέπει να ενισχυθούν. Ναι, Έχουμε μια αποστολή στο Μπασάρι Σαρίφ που είναι το φέουδο του Ντοστούν που είναι ένας εγκληματίας. Το ξέρουν όλοι. Ξέρουν ποιος είναι. Ποιος είναι λοιπόν ένας εγκληματίας πολέμου συνομιλητής μας που ελέγχει και τον πόλεμο και τα ναρκωτικά. Ποιον θα έχουμε σαν συνομιλητή. Αυτόν υποχρεωτικά πώς θα υπάρξει μια πραγματική συνεργασία στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία με ένα εγκληματία, γκάκστερ πρέπει να τον πω, ο στρατηγός του ε, Αυτό είναι οξύμορο, είναι μια καθαρή εσωτερική αντίφαση αυτή. Δεύτερο, τον Παμακό στο Μαλί. Τι κάνουμε, στέλνουμε στρατεύματα εκεί και μετά έχουμε τα προβλήματα. Ουσιαστικά εκεί ποια είναι, η ζάχαρη και το νερό. Δεν μπορούμε να πάμε στο βορρά λένε. Μα εκεί ακριβώς πρέπει να πάμε. Εκεί, στο Κιδάλ, στο Εντανίου, το Μπουκτού, εδώ και εκεί. Εκεί ακριβώς που υποφέρει ο κόσμος, τι γίνεται. Λαμβάνουμε υπόψη μας ε, ότι για να ελεγχθεί αυτή η περιοχή που είναι οι Ισλαμιστές, ε, οι εξτρεμιστές, ε, εκεί που γνωρίζουν τα μέρη, οι Τουάρεγκ είναι, οι Άραβιες είναι εκεί και ότι υπάρχουν μονάδες μάχημες. Ε, εκεί ακριβώς από αυτές τις φυλές γνωρίζουν τον τόπο και όχι οι νότιες φυλές. Για ποιο λόγο ακριβώς αυτό το διαλυμένο στράτευμα όχι από τον ε, βορρά αλλά από τον νότο θα πρέπει να επέμβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Καστάλντο μάλλον. Ε, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανάλυση σας. Μερικά πράγματα για ορισμένε αποστολές που μας εξηγήσετε. Το κοσυφοπέδιο. Και χθες ε, στη συνάντηση με χώρες αυτές ε, από λέει εδώ ακριβώς ε, έχουμε μια πληγή, ένα εμπόδιο. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα για την μελλοντική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ιστορική αναγκαιότητα. Δυστυχώς τι διαπιστώνουμε ότι εκεί ακριβώς σημαίνεται αυτό το σκάνδαλο πολλές και βαριές κατηγορίες από τον τόπιο τύφο σχετικά με αυτούς που στείλαμε εκεί και μιλάμε για τη μεγαλύτερη αποστολή και σαν προϋπολογισμό, σαν χρήματα, σαν άτομα που πήγαν εκεί. 1600 πήγαν και ο Μόγκερ, ε, ο πρώτος ορμοστής, έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι είναι στρατηγική περιοχή και ότι θα πρέπει να δούμε και ο επικεφαλής της αποστολής, νομίζω ότι και εκείνος είναι Ιταλός, είπε ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή απέναντι σε περιπτώσεις διαφθοράς. Πέστε μας λοιπόν, τα τελευταία νέα ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα και πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έτσι συγκεκριμένα, πώς θα μπορούσαμε να διορθώσουμε την εικόνα αυτής της αποστολής που αφισβητήθηκε τόσο και για την Παλαιστίνη. Απόλυτα συμφωνώ με όσα είπε Αφρονάρτ ε, για την αποστολή εκεί. Εδώ στη Ραφαν και στη Ραμάλα να σας πω κάτι. Αυτές τις μέρες τελευταίες θα το γνωρίζετε από τα θέματα που διαιρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αναγνώριση ή όχι της Παλαιστίνης. Πέρα από αυτό το θέμα, σωστό είναι ή όχι. Και εγώ το είπα και στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να δούμε, να αναγνωρίσουμε ένα κράτος χωρίς να του επιτρέπουμε ένα πραγματικό κράτος, δηλαδή μια πραγματική αποτελεσματική διοίκηση, μια αστυνομία, μια αξιόπιστη δικαιοσύνη. Σημαίνει ότι θα είμαστε υποκριτές και ότι θέλουμε να αποκρύψουμε την παλιότερη ευθύνη μας. Κατά την άποψή σας, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να διευρυθεί παραπάνω μετά από όσα διδαχτήκαμε αυτά τα τελευταία χρόνια για μια μελλοντική προοπτική, να πετύχουμε κάτι περισσότερο, για ένα πραγματικό Παλαιστινιακό κράτος που είναι αναγνωρισμένο από την εθνική κοινότητα, Μια είναι αξιόπιστη και η δράση του και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και ολοκληρώνω με την Λιβύη. Δεν είναι δική σας ευθύνη ότι δεν μπορούν να γίνουν και πολλά εκεί. Ξέρετε τα πλαίσια ότι είναι εντελώς αρνητικά. Βέβαια το να τρέφει κανείς αυταπάτες ότι μπορεί να ελέγξει χιλιάδες ε, χιλιόμετρα συνόρων, ακόμα και αν στείλουμε 100-200 άτομα εκεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αν ε, θα πρέπει να δούμε την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων. Θα πρέπει να το δούμε στρατηγικά ευρύτερα και με τον ήγερα την Αλγερία, την Αίγυπτο και την Τινησία ιδιαίτερα που βλέπουμε ότι Εκεί σημαίνεται ένα πέρασμα ιδιαίτερα θετικό, δημοκρατικό. Θα πρέπει να δούμε ένα νέο σύστημα, να μπορέσουμε να υπολογίσουμε και στις δικές τους ικανότητες, τη γνώση του εδάφους τους, γιατί ξέρουμε τα πράγματα αυτά. Κύριε Καστάλτα, σας παρακαλώ μήπως θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, μακρηγορώ, ναι. Λοιπόν, ναι, εάν δεν έχουμε γενικότερη εικόνα, δεν θα πετύχουμε τόσο εύκολα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κούκεν. Κύριε Πρόεδρε, ερωτώ. Το σκάνδαλο διαφθοράς Ιουλέξ. Θα το συζητήσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε παρακαλώ. Θέλω μια απάντηση για να ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω ή όχι επί του θέματος. Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Ωραία. Προκειμένου δύο ερωτήσει λοιπόν προς τον ε, εκλεκτό προσκεκλημένο μας. Ποια είναι εκτιμήσεις για το θέμα ότι ο κύριος Σοραϊλή έρευνα κατά πόσον η ΕΙΔΑ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διερευνήσει το σκάνδαλο και δεύτερον σχετικά με το θέμα τι λέμε στον πληθυσμό στο Κόσοβο τι κάνουμε από επικοινωνικής απόψεως για να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας τουλάχιστον. Και όλα Δύο ερωτήσει έχω. Η μία έχει τη Ράφα. Να το εξή. Η Χαμάς εξαπέλυσε 3.000 ρουκέτες κατά του Ισραήλ, κατά πολιτών και πιστεύω ότι θα ήταν μεροληπτικό να πούμε ότι το Ισραήλ μόνο προσπαθεί να καταστρέψει τη Γάζα. Δεύτερον, η κατάσταση προσομοιάζει με πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις μας στην περιοχή. Και με ποιο τρόπο και αν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με την ε, Γάζα, που μπορεί να ελέγχει την ε, Γάζα, αλλά οποία είναι αναγνωρισμένη στην τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, πώς συγκεράζουμε αυτά τα δύο. Τη στιγμή που υποτίθεται η Χάμά είναι και η εκλεγμένη αρχή, και η οποία όμω ακολουθεί το δρόμο τη επίθεση και τη τρομοκρατίας. Η κύρια ερώτησή μου θα ήταν μάλλον η εξή. Συζητήσαμε για πολυαριθμέ αποστολέ στο ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, γίνεται πολλής λόγος για την απόδοση αυτών των αποστολών. Όσον αφορά επίσης την πολιτική προμηθειών, θα επαναλήθουμε σε αυτό. Ακούω από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το ακούω και από άλλους, ότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίε υποτίθεται θα κρατήσουν ένα χρόνο, μετά από 6 μήνε δεν έχουν κάνει τίποτα γιατί η πολιτική προμηθειών είναι τόσο πολύπλοκη που τελικώ μετά από 6 μήνε δεν έχουμε τίποτα στη χέρια μα. Το εξοπλισμό και το προσωπικό έχει πάει επί τόπο, δεν κάνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αποστολών τη. Είμαστε παρκώ προετοιμασμένοι. Είναι δυνατόν να επιχειρήσουμε έτσι στο πεδίο από τη στιγμή που η πολιτική προμηθειών δεν αποδίδει. Πέρα από το οικονομικό θέμα και την γραφειοκρατία έχουμε ένα θέμα ασφάλειας του προσωπικού στην περιοχή που επιχειρεί χωρίς να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Όλερ. Άλλοι μιλητές. Όχι. Κύριε Κίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά όσον αφορά τα δημοσιονομικά, τον προϋπολογισμό μας. Για το 2004 ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΑ ήταν 314 εκατομμύρια. Από αυτά 299 αφιερώνονται στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΕΠΑ. Τα υπόλοιπα σε πρωτοβουλίες, σε μια εξάπλωση όπλων κλπ στο Μαλί μεταξύ άλλων που ξεκινάει τον Ιανουάριο να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε την αποστολή μέχρι τον Ιούνιο του 2015 συγκεκριμένα. Τώρα να προκύψουν και άλλες αποστολές το 2015 θα πρέπει να ξέρουμε και την ειδική εννοείται χρηματοδότηση για αυτές τις ξεχωριστές αποστολές. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι διευθυντές μου να εξεύρουν δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων. Εξετάζουμε πού μπορούμε παραλαμβάνω να εξοικονομήσουμε χρήματα χωρίς να φυγεί η εξοπιστία και η αποτελεσματικότητα των αποστολών μας. Θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί, θέλουμε οικονομίες, θέλουμε μια λιτή διαχείριση, δεν θέλουμε μεγάλε μεγάλες αποστολές. Έχουμε τις περιορισμούς μας εννοείται. στην Γεωργία για παράδειγμα έχουμε προσωπικό που είναι εκεί από το 2008 και μπορούμε να πάρει το σήμερα και αυτό θα κάνουμε και για όλες τις άλλες αποστολές κάθε φορά λέει θα ερωτούμε χρειάζεται οπωσδήποτε ο α ή ο β στην περιοχή και μετά αυτά θα τα υποβάλουμε στα κράτη-μέλη στο αμέσως προσεχές μέλλον για το Κίεβο δεν έχουμε παρουσία εκτός του Κιέβου αυτή τη στιγμή και λόγω ε, ασφαλείας όλα τα κρατημέλη θέλουν να περιοριστούμε στο Κίεβο. Υπάρχει βέβαια ένα στοιχείο το οποίο ήταν και στο Ρουγκάνς και το οποίο έχει αποσύρθει. Έχω αποσυρθεί από διάφορες περιοχές της ε, Ουκρανίας το Ντονμπάς ε, για παράδειγμα θα ξανούμε το θέμα πάντως η αποστολή αυτή τη στιγμή της ε, ΚΕΠΑ δεν θα επιχειρεί έξω από το Κίεβο τώρα για την ταχύα αντίδραση στην Γεωργία η αποστολή έχει στόχο την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων καμία σχέση με αντίδραση. Είναι θέμα βεβαίω τη ε, ΚΕΠΑ, εάν προκύψει τέτοιο ζήτημα, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για ένα σύστημα εγκαίρου προειδοποίησεω και τίποτα άλλο. Το θέμα είναι να επαληθεύσουμε αυτέ τις φήμες και πληροφορίες για συγκέντρωση ρωσικών δυναμίων στα σύνορα. Μιλάμε με του Ρώσους, έχουμε μια αμεσή γραμμή με την Οσυντία και την Απχαζία και μας λένε διάφορα πράγματα, εμεί δεν μπορούμε να μεταπιστέψουμε αλλά και η Γεωργία έχει ένα μνημόνιο συνεργασίας βάσει του οποίου δεν θα συγκεντρωθούν γεωργιανά στρατεύματα στα σύνορα στο πλαίσιο τη ρυθμή συμφωνία. Πρόκειται λοιπόν για ένα μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση και μόνο και τίποτα άλλο. Τώρα, για το ερώτημα όσον αφορά τη Ράφα και γιατί είμαστε καν στη ράφα. Είναι υγιής αυτός ο διάλογος, αν θέλετε. Τα κρατημέλη είναι διηρημένα επ' αυτού. Τρία-τέσσερα κρατημέλη λένε απλώς ότι η αποστολή πρέπει να παραμείνει επιτόπου για να προστατεύσει τον τοπικό πληθυσμό και να παραμείνει και το 15 βάσει συμφωνίας που έχουμε με του Παλαιστινίου. Χρειάζεται ένα τρίτος παρατηρητή η Παλαιστινιακή Αρχή μας θέλει εκεί γιατί είμαστε από τους ελάχιστους διεθνείς παράγοντες στην περιοχή βάση συμφωνίας. Είναι συμφωνία που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως όντως τελεί ενυπνώσει αυτή η αποστολή. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αν θέλετε και τα γραφεία είναι στο Τελαβίβ. Κάποια κρατημέλη πάντως βλέπουμε την αποστολή αυτή ως ακρογωνίο ε, λίθο κάθε μελλοντικής μας παρουσία στην Γάζα. Από εκεί πέρα ακολουθούμε τι εντολέ που έχουν ήδη δοθεί. Στο Αφγανιστάν η αστυνομία είναι δύσκολη. Γι' αυτό και συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο Μαζάρα Λισαρίφ και στην Καμπούλ. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά αν δεν ήμασταν εκεί τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Κανεί δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ότι δεν είναι σε επαφή ούτε με πολεμάρχους, ούτε με διαφέρμένου ούτε με εγκληματίε, Αλλά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολα. Έχουμε να κάνουμε ένα προβληματικό παρελθόν στη χώρα αυτή. Σίγουρα δεν εθαρρύνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή με ανθρώπου που εκ των πραγμάτων ε, είναι γνωστό ότι είναι εγκληματίε. Στον Παμακό τώρα και το Μαλί και πάλι με μια μη στρατιωτική αποστολή υπό τις διαταγές των κρατών μελών. Η κατάληξη, η κατάσταση με είναι αυτή που είπατε. Η αποστολή μας δεν έχει ως αντικείμενο να δώσει τέλος στον πόλεμο. Οι Γάλλοι έχουν και ισχυρή παρουσία, δρούν διμερός Η UTM πάντως ε, η δική μας δύναμη έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων του Μαλή. Από εκεί πέρα το Μαλή πρέπει να δημιουργήσει μια αξιόπιστη ισχυρή στρατιωτική δύναμη ασφαλείας. Εμείς απλώς έχουμε αυτή την πολιτική να υποστηρίξουμε την μη στρατιωτική αποστολή και βεβαίως τις μεταρρυθμίσεις ώστε κάποια στιγμή να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση και, τον, και της κυβέρνησης και του στρατού. Το Γιούλεξ Κόσοβο. Άκουσα δύο ερωτήσει. Πονήθηκαν διάφορα πράγματα, υπάρχουν φήμε, όντω. Δυσάρεστα είναι όλα αυτά, αλλά τα παίρνουμε στα σοβαρά και είπα ότι εκπρόσωπο στο δικό τη επίπεδο έχει κατά παράληψη δηλώσει ότι οι φήμες αυτές πρέπει να διερευνηθούν με διαφάνεια. Αν κάποιοι έκαναν κάτι πρέπει να οδηγηθούν ενώπιν της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Συνεχίζεται η έρευνα πάντως μετά από τις καταγγελίες μιας κυρίας το 2013. Αυτή η διερεύνηση οδήγησε στην μερική άρση ασυλίας κάποιων ε, στελεχών της αποστολής οι οποίοι τον οποίο η εντολή έφτασε στο τέλος της. Έχει αναλάβει η Ιντερπολ και διάφορες χώρες. Η διερεύνηση συνεχίζεται, για ευνότητες λόγους δεν μπορώ να σχολιάσω. Πάντως συνεχίζεται, παραλαμβάνω η διερεύνηση και σίγουρα θα φτάσουμε ως το κόκαλο. Η διερεύνηση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, παραλαμβάνω δεν στα χέρια μου, είναι στα χέρια της πάτης εκπροσώπου που είναι για την αποστολή. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο την ε, ικανοποιητική διεκπαιρέωση και ολοκλήρωση αυτής της διερεύνησης. Ε, πρόκειται για αποστολή στον τομέα του κράτου δικαίου και πρέπει να είναι λευκή ω περιστερά. Παραλαμβάνω ότι αν κάτι έχει στραβώσει βεβαίω θα το διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι να μην υπονομεύσουμε την αποτελεσματικότητα τη δράση. Έχω μιλήσει με υψηλά ισταμένους συναδέλφου και όλοι είναι υπέρ μια ταχεία ολοκλήρωσης της ανάκρισης και τη εν γέννη διερεύνησης. Η υπέτη έχει ορίσει τον κύριο Ζαν Πολσακέ, ο οποίο θα πάει επί τόπου πέντε μέρε, 14 Δεκεμβρίου, για να συνεχίσει τη διερεύνηση. Έχει εμφανιστεί και ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ε, και θα ξαναρθεί αρχές ή τέλη Ιανουαρίου να μιλήσει. Πάντως ε, έχουμε τέσσερις μήνες μέχρι τον Μάρτιο να ολοκληρώσουμε την έκθεση. Θα είναι δημόσια αυτή και είναι κάτι το οποίο φορά όχι μόνο το κόσμο αλλά και γενικότερα την εξοπιστία μας. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουμε την εξοπιστία της συγκεκριμένη αποστολή. Είπατε εκπρόσωπος ε, επαναλαμβάνω υποστηρίζει την διερεύνηση, δεν μπορεί να την επιταχύνει γιατί ακολουθούμε συγκεκριμένα ε, βήματα, αλλά να μην έχετε καμία εμβολία, θα διελευκάνουμε την υπόθεση και θα μάθουμε το μάθημα μας και τα μαθήματα αυτά θα τα εφαρμόσουμε αμέσως ε, παντού. Επαναλαμβάνω, είπε ότι εκπρόσωπος ε, είναι προσυλλομένη και έχει δεσμευθεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση αυτή. Ελπίζουμε να διευσεστούν οι φήμε, αλλά αν επαληθευθούν οι αρμόδιε αρχέ, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έναντι ουδήποτε υπευθύνου. Λιβύη. Κατάλαβα αυτό που είπατε για την περιφερειακή προσέγγιση. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. όντω. υπάρχουν εκατοντάδε, ανά χιλιάδε χιλιόμετρων συνόρων. Είναι και άλλες κυβερνήσει όμω στην περιοχή και άλλες χώρες το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο και έχετε δίκιο και συμφωνώ και περισσότερο πιστεύω υπάρχει μια περιφερειακή πτυχή δεν είναι μόνο η Λιβύη αλλά εξαρτάται πια από τα κρατημέλη και την ερώτηση κ. Όλε για το μέλλον μας στη Ράφα στη Ράφα ή οπουδήποτε κοντά στην Γάζα δεν θα συνεχιστούν εάν δεν εκπληρωθούν κάποια κριτήρια. Και για, για την μόνιμη παρουσία μας στη Γάζα εμείς θέλουμε να μιλάμε με την Παλαιστινική Αρχή και όχι με την Χαμάς. Μόνο όταν επανελθεί η Παλαιστινική Αρχή, μόνο όταν επανελέγξει την Γάζα, τη λωρίδα της Γάζας, τότε θα επανέλθουμε και εμείς, αλλά δεν μιλάμε με τη Χαμάς. Έχει σημειωθεί πρόοδος, όχι όσοι θα θέλαμε. Όμως επαναλαμβάνω, η αποστολή αυτή δεν θα επαναδραστηριοποιηθεί αν δεν επανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή. Εμείς ξεκίνησαμε την παρουσία μας εκεί το 2005 με την Παλαιστινιακή Αρχή Έχουμε και έναν εξάρτητο παρατηρητή. Ε, καλό είναι να εμπλεκεί και η Αίγυπτος ώστε να είναι τριμερής η αποδοχή της παρουσίας μας εκεί. Εμείς είμαστε ένας από τους πυλώνες. Υπάρχει μια πτυχή ασφάλειας, διότι πολλές φορές έχουμε ανοιχτές πολεμικές συγκρούσεις, στην περιοχή. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι να βρεθούν μεταξύ διασταυρωμένων πυρών, και το οποίο δεν το θέλουμε. Επίσης έχουμε τα σημεία διέλευση, τα συνοριακά σημεία. Όπως και στην ε, Γεωργία δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του προβλήματος, δεν θέλουμε να είμαστε στην περιοχή των ενόπλων σειράξεων. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή ε, η αποστολή αυτή θα γίνει ξανά ειρηνευτική αποστολή. Τώρα για το Κόσοβο και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Εντοπίστηκαν προβλήματα όντω οικονομικά στι προμήθειε, τη κ. Σόλερ. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα όλων των αποστολών. Όντω Όντως 7, 8, 9 μήνε πολλέ φορέ για μια αποστολή να προμηθευτεί αυτά που χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ ο χρόνο. Και είναι λίγο παράδοξο, γιατί υποτίθεται να πηγαίνουμε εκεί για να υποστηρίξουμε γρήγορα κάποιε κυβερνήσει. Το Δεκέμβριο του 2013, στην σχετική παράγραφο, στη συμπεράσματα του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλεί την υπατή εκπρόσωπο, τον τότε μάλλον υπατή εκπρόσωπο, να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Περιμένουμε τώρα από την ΕΙΕΔ να κάνει την πορεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2015 ελπίζω ότι θα το έχουμε ολοκληρώσει. Όντω ο δημοσιονομικό κανονισμό πάντω δεν είναι ευέλικτο. Εγώ θα ξανάγραφα κάποια άρθρα, αν θέλετε, για να μπορούμε να μυθευόμαστε αυτά που χρειαζόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να τηρηθούν φυσικά και οι αρχές της ορθής οικονομικής διαχείρισης και να διευκολύνουμε και τους ελέγχους. Τα πράγματα πάντως έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα. Όντως κάτι πρέπει να αλλάξει για να επιταχύνουμε τις σχετικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Κίν, θέλετε την καλοσύνη να μας πείτε δύο λόγια ακόμα για την αποστολή στη Γεωργία και τις πρακτικές δυνατότητες που έχετε για μια ισορροπημένη εκτέλεση των καθηκόντων σας και γενικά για την προσέγγιση σας στο θέμα της Οσετίας, της Νότιας, της νότιας Οσετίας, της Απχαζίας και την ανάγκη να εξασφαλιστούν σαφείς ορισμοί ώστε να παρακολουθείτε την κατάσταση εκεί, γιατί ξέρουμε ότι η Ρωσία δεν είναι διτεθειμένη να συνεργαστεί. Μιλάτε για μια ουδετερή ζώνη. Η Ρωσία ξέρουμε ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του 2008, τη συμφωνία μεταξύ Μετβέτεφ και Σαρκοζή. Άρα τι σχέδιο έχετε, πώς θα θέλατε να παρακολουθείτε την κατάσταση και να ενημερώνετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και νωρίτερα, ο καθένας, μόνο αυτό που έχουμε δει, αυτό που ξέρουμε μπορούμε να αξιολογήσουμε. Αυτός ο μηχανισμός άμεσης ε, ανταπόκρισης στην Απχασία μπορεί να στηριχθεί μόνο στις θέσεις και τις απαντήσεις των Ρώσων. Και από την άλλη είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώνουμε ερωτήματα με βάση τις φήμες που ακούγονται και τις ε, αναφορές. Έστω και φιλικά δηλαδή, πάντως υπάρχουν φήμες ότι συγκεντρώνονται όπλα, από την πλευρά της, της Απχασίας ότι είναι δορυφόρο ή πάνω στην περιοχή και μπορεί μεν εμείς να μην είμαστε σε θέση να το ε, επαληθεύσουμε αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές τις αναφορές. Υπάρχουν επίσης περιπολίες διαρκής όλη τη βδομάδα, όλη τη μέρα ίσως όχι πάντα μέσα στη νύχτα, αλλά διαρκής μέσα στην εβδομάδα. Περνάει ο κόσμος στα σύνορα, μιλάει και άρα προσπαθούμε και εμείς από πλευράς μας να δούμε αν μπορούμε να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε τουλάχιστον από την πλευρά τη γεωργική όπου βρισκόμαστε ε, τι είδους ανάπτυξη και έκταση στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμών υπάρχει από την άλλη στην Απχαζία. Ευχαριστώ θερμά. Πολύ καλό το τελευταίο αυτό σημείο ως εισαγωγή στο επόμενο θέμα μας. Γνωμοδότηση Έλλαρ. Είναι εισηγητής ο κύριος Έλερ για θέματα που αφορούν ε, δημοσιονομικούς κανόνες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο να εξασφαλιστεί περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη δράση. Κύριε κύριε ευχαριστούμε θερμά. Το θέμα αυτό θα παραμείνει παγίως στο πρόγραμμα των εργασιών μας. Θα παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση και στο βαθμό του δυνατού θα σας καλούμε για τα λέγια απόψε. Ευχαριστώ πολύ και έκλεισε το θέμα αυτό. Thank you. Now we... Ευχαριστώ. Σα Σας φέρω το επόμενο σημείο της ημερήσια μας διάταξη. Έλερ, ο εισηγητή και με τους κυρίους εισηγητές έχουν το λόγο από τις πολιτικές ομάδες ε, και μετά για περαιτέρω συζήτηση και θα ψηφίσουμε στην συνάντησή της Πότε θα γίνει αυτό τον Ιανουάριο, ναι τον Ιανουάριο. Και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι το Δεκέμβριο 10 του μήνα μέχρι το μεσημέρι. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, εντάξει σημειώστε τα αυτά. Κύριε Έλλερ, ο λόγος σε εσά. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί μπορεί να προσδιορίσει τη θέση, τη στάση της Επιτροπής μας. Ε, είχαμε στο παρελθόν συμβολικά περισσότερο και πολιτικά ζητήματα με, με, με συμβολικά και πολιτικά ζητήματα να ασχοληθεί, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει μεγάλη και κρίσιμη σημασία γιατί μπορούμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση προς το θέμα αυτό που δεν είναι μια γνωμοδότηση μόνο. Βέβαια, εγώ επέλεξα τη μορφή της γνωμοδότηση γιατί θα μα επιτρέψει να συζητήσουμε όπω και στο παρελθόν το τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρακτικά στην ουσία, τι είδου συμβολή μπορεί να προσφέρει η δική μα Επιτροπή σε σχέση με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, νομίζω ότι θα μπορέσω να σας πείσω για τη σημασία των θεμάτων αυτών και, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΑ. Της ΚΕΠ, μάλλον. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν παρουσίασε νέες προτάσεις ευθυγραμμισμένες στον δημοσιονομικό κανονισμό με τις διατάξεις των νέων οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες με προτάσεις οι οποίες αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία να ενσωματώσουμε μια τροποποίηση του άρθρου 190 με τις ε, ε, προμήθειες για εξωτερικές δράσεις και έτσι να αντιμετωπίσουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Πρόκειται για κανόνες οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ε, και επάχρηματοδοτούνται από τον νέο προϋπολογισμό και είναι περίπλοκοι. Η γενική κανονισμοί αυτοί για τις προμήθειες δεν μπορούν να ισχύουν και στην ΚΕΠΑ και την υποχρέωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις των γενικών ε, ε, οι γενικές διατάξεις για τις προμήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε ε, τεράστιες καθυστερήσεις, σκανδαλωδώς τεράστιες καθυστερήσεις και ουσιαστική αποδυνάμωση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα πρέπει οι αποστολές αυτές να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον κρίσεως και μέσα σε μια χρονική περίοδο περιορισμένη ξεκινούν με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου που αναγνωρίζει ότι χρειάζεται κατεπίγουσα ανταπόκριση σε μια κρίση. Παρ' όλα αυτά οι φυστάμενοι κανόνες, οι δημοσιονομικοί κανόνες προσδιορίζονται ε, έχουν προσδοριστεί μάλλον για μια λειτουργούσα εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και όχι για κρίσεις, ε, περιοχές και καταστάσεις κρίσης όπως το Μαλί ή το Νότιο Σουδάν και, όπου χρεια... και συχνά χρειάζεται να περάσουν και έξι μήνες για να ληφθεί μια απόφαση πάνω σε ένα διαγωνισμό. Εδώ λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη να πηγαίνετε λίγο πιο αργά. Παραδείγματα τα οποία για μένα είναι έως και τραγικά και δείχνουν πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τις αποστολές μας. Ας πούμε, ελικοδρόμιο, 50.000 δολαρίων κόστους. Εάν χρειαστεί 6 μήνες για να υλοποιηθεί, για να προχωρήσει, ουσιαστικά εξετερώνει την αποτελεσματικότητα μιας αποστολής που έχει διάρκεια ενός έτους. Εάν πρέπει να κάνουμε προμήθειες ε, ε, πετρελαίου στη Γεωργία, με δημόσια και διεθνή, με δημόσιο και διεθνή διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου στη Γεωργία. Χάνουμε κάθε αποτελεσματικότητα. Έχει συμβεί αυτό. Χρειάστηκαν εννέα μήνες για να ολοκληρωθεί ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός και πολλά άλλα παραδείγματα μπορώ να σας φέρω προς την κατεύθυνση αυτή. Και έτσι φτάνουμε μέχρι το σημείο να θέτουμε σε κίνδυνο και την ίδια την ασφάλεια του πολιτικού προσωπικού που έχουμε είτε πρόκειται για αποστολές κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων και δεν έχουν παραδείγματι μέσα επικοινωνίας και χρησιμοποιεί ο καθένα το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσει, πρέπει να κοιτάξουμε σε ποιο βαθμό μέχρι και θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων που στέλνουμε σε αυτές τις χώρες. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι συμφωνούμε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να καθυστερούμε την ανάπτυξη του δυναμικού κατά μισό έτο, περιμένοντα να γίνουν αυτοί οι διεθνεί διαγωνισμοί. Η τροποποίηση λοιπόν και η γνωμοδότηση, γιατί όπω είπα δεν είναι απλώ γνωμοδότηση, είμαστε σε διαρκή και άμεση επαφή με του συνάδελφου από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο αυτό άρθρο θα πρέπει να ενταχθεί και να σημάνει με την τροποποίηση αυτή Άλλωστε, σε ευθεία γραμμή και με τι αποφάσει του 2011 του Συμβουλίου, να λέει λοιπόν το άρθρο αυτό με τροποποίηση ότι θα εξασφαλίσουν οι κανόνες, ε, ε, θα συμπεριλαμβάνουν ειδικέ διατάξεις για την ε, προμήθεια υλικού που χρειάζεται για τις αποστολές υπό την ΚΕΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστούν η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η εγκατάσταση ιδιαίτερως των κατάλληλων και ταχείων διαδικασιών και το καθεξής. Εδώ αυτό που λέμε πάνω απ' όλα δεν είναι ότι ζητούμε παρέκκληση από τους υφιστάμενους κανόνες. Εγώ βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει μια κατεξουσιοδότηση πράξη περισσότερο και είμαστε σε ευθεία γραμμή ε, με τους συναδέλφους της Επιτροπής των Προϋπολογισμών ως προς το θέμα αυτό για να δούμε πώς θα το διατυπώσουμε και πώς θα το διατυπώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Άρα θέλουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο άρθρο για τις ε, αποστολές της ΚΕΠΑ και αναλόγως να προχωρούμε με κατεξουσιοδότηση πράξη. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και άλλες διατάξεις των δημοσιονομικών κανονισμών, το, οι οποίες τροποποιούμενες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας αποστολών. Οι εφαρμοστικές εξουσίες, για παραδείγματι, θα μπορούσαν να εκχωρηθούν στον διοικητή ή τον επικεφαλή της πολιτικής αποστολή. Δεν εισάγω όμως τώρα αυτήν την ε, τροποποίηση, σεβόμενο το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά καλώ την Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και με την παρουσίαση μιας προτάσεως να μας ε, προτείνει αυτή την τροποποίηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό πάλι πολύ βραδύ που δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να συμφωνήσετε με την γνωμοδότηση αυτή η οποία δεν είναι ακριβώς ε, γνωμοδότηση είναι μια συζήτηση embedded, ενσωματωμένη στην διαδικασία της Επιτροπής των Προϋπολογισμών και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έλερ και τώρα παρακαλώ τους σκυλιώδεις εισηγητές να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Φερνάρτες Άλβαρες, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Συγχαρτήρια στον εισηγητή Έλερ για αυτή την εργασία του αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και τις επόμενες εβδομάδες θα εργαστούμε επίσης εντατικά και θα πετύχουμε μια συμφωνία στην Επιτροπή. Σαν μέλος της Επιτροπής εδώ, εδώ και μερικούς μήνες πρώτη μου είδα τις δυσκολίες για πολλές ευρωπαϊκές αποστολές επιτόπου και ακούσαμε εδώ στην Επιτροπή παρεμβάσεις από εκπροσώπους ενόπλων δυνάμεων σε διάφορες ε, δράσεις στην Αφρική και παρατηρήσαμε να σημειώσονται προβλήματα όσον αφορά την ταχύτητα των παρεβάσεων αυτών και σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να παρακάμψει πολλά εμπόδια από αυτά που συναντάμε στις αποστολές μας. Η σοσιαλιστική ομάδα συμμερίζεται την ε, άποψη αυτή ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα για τις ευρωπαϊκές αποστολές με μηχανισμούς ε, συντονισμού ανάμεσα στις ε, στρατιωτικές δυνάμεις των διαφόρων κρατών, τα στρατιωτικά σώματα των κρατών μελών και μια στρατηγική και μια βιομηχανία μπορούμε να πούμε άμυνα στην Ευρώπη και να μπορέσει να βοηθηθούν και τα εργοστάσια, οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις, το σύνολο της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Σχετικά με τον κανονισμό που μας απασχολεί, να σας πω ότι συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη ότι το 190 άρθρο θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί για μια παρέμβαση πιο ευλίγιστη για τα διάφορα σχέδια και να έχουμε υψηλότερη ταχύτητα στις ε, συναντήσεις μας, στις επαφές μας όπως είπαμε και προηγουμένως είναι πολύ θετικό για να βελτιώσουμε αυτούς τους μηχανισμούς με ευληγησία για λήψη απόφασης και επιτόπου και επίσης θεωρούμε ιδιαίτερα θετική την ε, μεταρρύθμιση, την αθεώρηση αυτού του 190 άρθρου και τις επόμενες εβδομάδες για να διευκολύνουμε την εργασία για τα στρατεύματα αυτά, στρατικές αυτές δυνάμεις και επαναλαμβάνουμε ευκαμψία και ευληγησία και είμαστε πεπισμένοι ότι εδώ το Κοινοβούλιο και οι επιτροπή μας θα λάβουν και τους επόμενους μήνες τις κατάλληλες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Ε, Κυρία Πρόεδρε, το το συζητάμε είναι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε κανόνες σε όλα τα πράγματα. Από την πλευρά μου με ενισχύει το θέμα και η ομάδα μου, η πολιτική μου ομάδα ανησυχεί το θέμα της συμπληματικότητας των ενεργειών μας με τον ΝΑΤΟ. Και η ΕΦΕΤ το ίδιο έχει πει. Πρέπει να υπάρχει συμπληματικότητα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δράσεις αυτές. Θέλει προσοχή το θέμα, θέλουν περαιτέρω εξέταση οι δράσεις μας. Ερωτώ όμως, το μέγεθο των δρασιών μας δικαιολογεί όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχουμε κανόνες σύμφωνοι αλλά να προστατεύουμε μεταξύ άλλων και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια αναλογικότητα ας πούμε στο μέλλον θα εμπλέκονται παρκώς οι δυνάμεις μας η αμυντική βιομηχανία έχει νόημα το όλο πράγμα και θα αναλαμβάνουμε δράσεις που έχουν νόημα γιατί προς το παρόν έχουμε παρουσία σε πολύ μικρή κλίμακα που είτε είναι μελιτέα είτε περιφερειακού χαρακτήρα. Δηλαδή ασχολούμαστε μόνο με, την, με τις περιφέρειες στην άμεση γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή λοιπόν οι κανόνες, αλλά θα κάνουμε κάτι το οποίο να έχει και νόημα σε επαρκή κλίμακα. Και αν ναι, τότε πρέπει να βρούμε και τις κατάλληλες μεθόδους και μηχανισμούς για να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας. Και εκεί μπαίνει το θέμα Τη ευελιξία των κανόνων. Μήπω τότε θα χρειαστούμε διαφορετικούς κανόνες. Δεν θέλω να βρεθούμε εν κενό που οι σχετικά με τα οικονομικά θα λαμβάνονται με τρόπο αυθαίρετο και χωρίς να συνάδουμε κανένα κριτήριο. Το θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό παρακαλώ. Κύριε Σάντος. Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους των φιλελευθέρων, σύμφωνα με την ανάγκη αλλαγών εδώ, του 100 και του 109, υποστηρίζω επίση την τροπολογία της ΑΦΕΤ, πρέπει οι προτάσεις να είναι ευλογέ, να συνάδουν με τους ε, λογιστικούς οικονομικούς κανόνες, να ικανοποιούν το ελεγκτικό συνέδριο, το είπε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό και εννοείται όλα να συνάδουν με το επεξηματικό σημείωμα αυτής της πρότασης ψηφίσματος. Εκ μέρους της ΑΛΤΕ ε, υποστηρίζω λοιπόν την ε, άποψη αυτή. Κύριε Λέση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά με την αδειά σας. Συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Έλερ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θα ήθελα ξεκινώντα να κάνω μια βασική τοποθέτηση. Λυπούμε ιδιαίτερω για το ότι οι σημαντικές συζητήσεις της Επιτροπής μας, της Επιτροπής ε, Θεμάτων Αμήνη, ε, διεξάγονται με άδεια έδρανα. Λυπούμε πολύ για το της προοπτικής εξέλιξης αυτής της Επιτροπής και των συνεδριάσεών της. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε με τους συντονιστές εάν φταίει η θεματολογία που επιλέγεται, εάν τυχόν συμπίπτουν αυτές οι συνεδριάσεις συχνά και με άλλες επιτροπές. Πάντως είναι πολύ κακές αυτές οι επιδόσεις ως προς την παρουσία των συναδέλφων στην Επιτροπή. Για το σημείο λοιπόν αυτό. Έχουμε όντως να κάνουμε με πολύ σοβαρές ε, και κατά βάση εκτιμήσεις, θεμελιώδεις εκτιμήσεις που έχουμε ξανασυζητήσει σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής μας σε σχέση με τον προϋπολογισμό για την έρευνα ιδιαίτερος και δει τον προϋπολογισμό που, να που αφορά την έρευνα με πιθανή στρατιωτική χρήση. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση τροπολογίας της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων, ιδιαίτερα στο σημείο που αναφέρεται το «to be applied in all CSDP missions», να, να εφαρμόζεται σε όλες τις αποστολές και πα. Δηλαδή όλε τις αποστολές με στρατιωτικό χαρακτήρα, κατά κύριο λόγο, λέει ο μιλήτρια. Κύριος Έλλερ, όχι, όχι, όχι, να σας διακόψω το τυπικό κομμάτι, το στρατιωτικό, δεν χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ω εκ τούτου δεν υπάρχει αναφορά σε στρατιωτικέ δαπάνε. Πρόκειται για πολιτικό κομμάτι τη ΣΚΕΠΑ. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Ε, η Πρόεδρος. Σας παρακαλώ μην αρχίζουμε τους διαλόγους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε τι απαντήσει στη συνέχεια. Κύριε Λόζινγκ, ναι, Καλά, παρόλα αυτά, χαίρομαι που κάνατε αυτή τη διευκρίνηση σύντομα κύριε Έλερ. Πάντως πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία όπως έχει δεν είναι τόσο σαφής όσο αυτό που είπατε. Εγώ ερμηνεύοντας το κείμενο που διαβάζω καταλαβαίνω ότι αφορά αποστολές χαρακτήρα στρατιωτικού. Και άρα θα ήθελα πολύ ξεκάθαρα να υπάρξει αναφορά στο άρθρο θα ήθελα να κάνω την παραπομπή στο άρθρο 41 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λέγεται ότι οι δαπάνες ε, για τη λειτουργία του οργάνου προκύπτει από την ε, διατύπωση του παρόντος άρθρου και οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από το κεφάλαιο αυτό ε, χρηματοδοτικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη εξαιρέσει των στρατιωτικών δαπανών, δαπανών που έχουν να κάνουν με στρατιωτικέ και αμυντικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνε επιβαρύνουν τα κράτη-μέλη με βάση την κλίδα κατανομή επί του ΑΕΠ και τα κράτη-μέλη δεν δεσμεύονται, δεν υποχρεούνται δεν μπορούν να υποχρεωθούν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δαπάνες. Γιατί κύριε Έλερ, το εξηγήσατε εσείς τώρα. Έτσι λοιπόν πρέπει να διευκρινιστεί και μέσα στο κείμενο. Η διατύπωση της ε, τροπολογίας για μένα οδηγεί, γιατί για μας, για, ε, για μας λοιπόν δεν είναι συμβατή με τη συνθήκη. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ πολύ. Έχω αναλάβει σκιώδης εκ μέρους των Πρασίνων για την έκθεση αυτή. Αισθάνομαι λίγο σαν το Φρανκ Σινάτρα και το τραγούδι The Shadow of a Smile. Σκιώδης, λοιπόν, για τα πάντα. Ε, συμφωνούμε με αυτά που ο κύριο Σέλλερ, ε, διαφωνούμε συγγνώμη για αυτά που είπε ο κύριο Σέλλερ, σχεδόν σε όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτές τις αποστολές της ε, ΚΕΠΑ ότι δεν λειτουργούν με βάση τις συνήθεις, ε, τους συνήθεις όρους της αγοράς. Μας έφερε κάποια παραδείγματα ο κύριος Έλερ, το ελικοδρόμιο και όλα αυτά τα γελία παραδείγματα. Όταν έχω επιχειρησιακή διοίκηση αναλάβει και χρειάζομαι έναν υπολογιστή, πρέπει να τον έχω τώρα στα χέρια μου, όχι σε δύο χρόνια και όντω μπορεί και να κοστίσει ανθρώπινε ζωές η καθυστέρηση. Πάντω σημειώνω μια σειρά από μικροπαρεξηγήσεις σε σχέση με το τι είναι η πολιτική πολιτικής χρήσης ε, προμήθειας και τι στρατιωτικής. Ίσως λοιπόν, ίσως να ήταν σκόπιμο να κάνω μια τροποποίηση στην πρότασή σας με την προστίκη του όρου civilian, πολιτικός. Για να είναι πολύ το σαφές το τι εννοούμε εδώ. και έτσι να είναι σαφές ότι αφορά τις πολιτικές αποστολές, μη στρατιωτικές αποστολές τη ΚΕΠΑ. Αυτό θα θέλω να σας προτείνω. Το μόνο. Και επίσης συμφωνώ με την κυρία Λούιζινγκ ότι είναι πονίδιστον το ότι είμαστε τόσο λίγοι εδώ. Αλλά και στην προηγούμενη θητεία θα ήθελα να πω ο, μάλλον το έχω ξαναπεί και στην προηγούμενη θητεία. Αφού είναι εδώ η κυρία Λέζινγκ, εγώ προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Καλώ λέει η πρόεδρο και σε ευχαριστώ. Οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Παραντή. Θέλετε κύριε Παραντή να λάβετε το λόγο για κάποια σχόλια και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή όλες τις ε, παρεμβάσεις των ε, κυρίων βουλευτών. Βεβαίως συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα να δρούν ταχαίως και αποτελεσματικά οι αποστολές μας στις διάφορες περιοχές. Θεωρούμε πάντως ότι πολλά ήδη έχουν ε, εξασφαλιστεί, η ευελιξία, αλλά και οι διαδικασίες που υφίστανται ήδη επιτρέπουν να δοθεί ταχεία ανταπόκριση με βάση τις ανάγκες μιας αποστολής. Φερρυπίν. Στους ισχύοντες κανόνες προβλέπεται ότι οι διαδικασίες για την προμήθεια, για τις προμήθειες, όταν υπάρχει κατάσταση κατεπίγουσα ή κρίσεως, είναι διαδικασίες κατόπιν διαπραγματεύσεως. Για τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς, με την ε, ανακήρυξη μιας καταστάσεως κρίσεως ή η διαπραγματεύσιμη διαδικασία ή η κατόπιν διαπραγματεύσεως διαδικασία αφορά μία μόνο διαδικασία διαγωνισμού. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Για το διοικητικό διαγωνισμό επίσης το ίδιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ε, προτάσεις στη διαπραγματεύση στην υποδιαπραγμάτευση διαδικασία. Εμεί προτείνουμε τώρα, με το κείμενο που εξετάζετε κι εσεί, να υπάρξει μόνο μία προσφορά. Αυτό λοιπόν με μια πολύ ειδική διαδικασία ε, κατόπιν διαπραγματεύσεως διαγωνισμών με μία μόνο προσφορά μας φαίνεται πολύ κατάλληλη. Επιπλέον έχουμε και στοιχεία ευελιξίας εγκαθιδρύση. Φερρυπίν. Προβλέπεται αποθήκη με τον πάγιο, παγιος αναγκαίο προϋπολογισμό για τις αποστολές. Είναι διαθέσιμος αυτός και υπάρχει όλο το βασικό υλικό. Οι υπολογιστές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, χάρη στην αποθήκη αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα τηλέφωνα, για τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά υφίστανται και είναι διαθέσιμα αμέσως, χάρη στην αποθήκη. Βέβαια κοιτάμε να δούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Επί παραδείγματι μιλάμε με το Συμβούλιο για την ανάπτυξη ενός κέντρου κοινών ε, υπηρεσιών Shared Service Center δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε σε σχέση με την ε, υποστήριξη που βλέπουμε από το Συμβούλιο για την αποστολή. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς δηλαδή με όλες τις αποστολές και πά. Μπορεί να είναι μια κεντροποιημένη υπηρεσία που θα μοιραστεί μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της επιτροπής ε, Ειδικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως ε, με ένα σύστημα συμβάσεων. Ένα σύστημα κοινών υπηρεσιών το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία, τη διαχείριση των πόρων και τις προμήθειες των αποστολών. Ήδη λοιπόν πολλά πράγματα έχουν γίνει και βεβαίως θέλουμε να κοιτάξουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που καταγράφονται και από τον εισηγητή κύριο Έλερ. Αυτά που μας είπε εγώ δεν τα γνώριζα για το ελικοδρόμιο, Φερρυπίν. Πάντως είμαστε έτοιμοι. Τα παρακολουθούμε με τους αρμόδιους ε, των Επιτροπών και την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης θα συζητούμε και θα προχωρήσουμε. Τώρα για να δώσω κάποιες απαντήσεις σε σχέση με το νομοθετικό πλέγμα που προτείνεται από την τροπολογία. Οι αποστολές έχουν βεβαίως δημοσιονομικά καθήκοντα, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε και τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, όπως ανέφερε και κάποιος βουλευτής. Έτσι λοιπόν, εάν εκχωρήσουμε δημοσιονομικά καθήκοντα για τους, προς τους εταίρους μας για τις αποστολές, επί παραδείγματι, θα πρέπει να περάσουν από μια λεγόμενη αξιολόγηση πυλώνα, pillar assessment, όπου προβλέπεται η αξιολόγηση των προμηθειών που χρησιμοποιούν, των διαδικασιών προμηθειών που αξιοποιούν. Ε, συνήθως θέλουμε να δίνουν ε, τα ίδια εχέγγυα αυτές οι διαδικασίες με τις δικές μας. Για τις αποστολές όμως έχουμε επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία. Ο δημοσιονομικός κανονισμός όπως είναι διατυπωμένος τώρα προβλέπει μια πιο μακρά περίοδο προσαρμογής της αξιολόγησης και την καθίδρυση των πυλώνων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προμήθειες. Και σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, πράγμα το οποίο ομολογώ πως διαπιστώνουμε για κάποιες από τις αποστολές, είναι υποχρεωμένη και δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα μέτρα τα οποία εν προκειμένου συνεπάγεται μία εκ των μια ετεροχρονισμένη, μια εκ των προτέρων ε, θεώρηση, αναδρομική μάλλον θεώρηση. Αλλά θα ήθελα να πω για τους κανόνες που προτείνεται εδώ, γιατί εντάξει ότι δεν θα χρειάζεται κατεξουσιδότηση συμπράξη. Αυτό ούτως ή άλλως προβλέπεται για υπηρεσίες αποκεντρωμένες και άλλους οργανισμούς με βάση τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αποτελεί τη, βασική, τη νομική βάση. Η ε, συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που αποτελεί τη νομική βάση για την ΚΕΠΑ και όχι η συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τι αποστολέ, να εγκαθιδρύσουμε, να υιοθετήσουμε δημοσιονομικού κανόνε, να μην προχωρήσουμε σε κατεξουδότηση πράξη. Πρέπει απλώ να υιοθετούμε δημοσιονομικού κανόνε και κάποιοι από αυτούς μπορεί ακόμα να μην έχουν υιοθετηθεί, αλλά εάν κομμάτι, αν εκχωρηθεί κομμάτι της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού στη συμφωνία αυτή εκχώρησης, ήδη έχουν γίνει προσδιοριστεί μια σειρά δημοσιονομικών κανόνων, που όμως ενδεχομένως για τις προμήθειες να χρειάζονται περαιτέρω συμπλήρωση και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να ετοιμάσει ένα πάγιο έντυπο, ένα υπόδειγμα για αυτούς ε, τους δημοσιονομικούς κανόνες που αφορούν τις προμήθειες. Προτείνουμε λοιπόν να ευθυγραμμιζόμαστε με τις αρχές που είναι πολύ γενικές, αφενός, αφετέρου να υπάρχει η συνέχεια της προμήθειας και δεν χρειάζονται νέα μέτρα σε σχέση με αυτά που έχουμε. Όταν χρειάζεται δίνουμε αναδρομική θεώρηση, έγκριση. Για την ε, ιδέα που ακούστηκε εδώ νωρίτερα από έναν από τους βουλευτές, ίσως να τον συγητής μάλιστα, με συγχωρείτε, για το θέμα του διοικητή της πολιτικής επιχείρησης, της μη επιχείρησης. Εδώ δεν είναι τροπολογία αυτό που προτείνεται, έχετε ωστόσο δίκιο που την προτείνετε διότι θα ήταν αντίθετο πιστεύουμε στο πλέγμα αρμόδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τις αρχές για την εφαρμογή, την εκτέλεση του προπολογισμού του άρθρου 137, δηλαδή ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να, να εκτελέσει τον ε, προϋπολογισμό. Επομένως, αν πρέπει να περάσουμε από έναν ε, ε, διοικητή μη στρατιωτικού προσωπικού που, είναι υπάλληλος, που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης ξεπερνάμε, αντιπαρερχόμαστε τις διατάξεις σχετικέ σχετικές με την εκτέλεση του προπολογισμού που μιλούν μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ελπίζω να απάντησα στα ερωτηματικά που προέκυψαν. Δεν χρειάζεται η τροπολογία, επανέρχομαι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Λειτουργούν ευελιξία υπάρχει. Συνεργαζόμαστε με αυτούς που καλούνται να υλοποιήσουν τις πολιτικές σε βαθμό παροχής και υποστήριξης και αρρωγής. Αλλά πάντως δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται η οδός των ε, κατεξουσιών συμπράξεων να επιλεγεί γιατί δεν θα είναι η σωστή δράση. Ευχαριστώ πολύ. Η, Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, παρακαλώ, ο κύριος Καλυμπίκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Για πέντε χρόνια εργάστηκα στις προκηρύξεις της Επιτροπής και οι εσωτερικοί κανονισμοί όλα αυτά τα θετικά και έχουμε και καθημερινά παραδείγματα σε αυτή την αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Μπορούμε να ταξιδεύουμε φτηνότερα, οι τηλεπικοινωνίες είναι φτηνότερες και μετά. Όταν έφτασα το ΕΣΕΕ, e, στη διόλη διαχείριση παρόμοιων ενεργειών, διαπίστωσα ότι οι σημερινοί κανόνες της αγοράς για τις εξωτερικές ενέργειες είναι ξεχωριστά, ξεχωριστές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τις προκηρύξεις διαγωνισμών και είπε μερικά παραδείγματα συγητής ε, ναι, και καθημερινής πραγματικότητας. Αυτά τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε στην Επιτροπή για περισσότερη ευληγησία και ευκαμψία των σημερινών κανόνων και μια προσαρμογή στις πραγματικές υπερχειρησιακές ανάγκες των αποστολών. Σήμερα, αν θέλουμε κάτι να προσφέρουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μετά από το τέλος της θητείας. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε μια δραστηριότητα οικονομική όπως το κάνουμε ας πούμε διοικητικά. Ε, αλλά θα πρέπει να το, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μια απόσταση 2-3 ετών. Σήμερα εργαζόμαστε στην περίπτωση κρίσεων, επαναλαμβάνω και για αποστολές, αλλά πολλές φορές ε, αυτή η έννοια περί κρίσης δεν λαμβάνει υπόψη οικονομικά. Αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί έτσι από τον ε, επικεφαλής ακριβώς την Επιτροπή που είναι και εκείνος που αποφασίζει για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια κάποια συμβατότητα. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδύσουμε τις ενέργειές μας. Τι βλέπουμε, Κωσυφοπέδια, Γεωργία και Αφγανιστάν θα μπορούσαν να, να ξεκινήσουν οι ε, ίδια αυτά μέρη με τις διαδικασίες αλλά αλλού χρειάζεται μια αξιότηση της Επιτροπής από τη στιγμή που θέλουν να προκηρύξουν ένα διαγωνισμό, μια, κήρυξουν μια πρόσκληση ενδιαφέροντας από τη στιγμή που το ποσό είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα με όσα εξήγησε ήδη ο εισηγητής πριν από λίγο και έτοιμος είμαι να δω από πώς θα υπάρξει η σχετική πρόοδος. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πω ότι εγώ για τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, τα είχα δει αυτά τα πράγματα από κοντά και νομίζω ότι τα παρακολουθεί και η Επιτροπή βλέπουμε το πώς εκφράζεται σχετικά πάντως αυτά είναι τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ σημαντικά πριν να δούμε από κοντά Να διευκρινίσω για άλλη μια φορά τα βασικά εδώ μιλάμε μόνο για τις μη στρατιωτικές αποστολές. Δεν υπάρχει καμιά πρόθεση επιλογής πολιτικής. Απλούστατα, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρηματοδοτεί στρατιωτικές αποστολές. Αυτές προκύπτουν από το μηχανισμό Αθηνά των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, και ως προς τις πολιτικές επιλογές, αλλά και ως προς την νομική βάση, η κατάσταση είναι σαφής και γι' αυτό η διατύπωση της τροπολογίας. Τώρα ίσως θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι πρόκειται για πολιτικές αποστολές, άλλωστε το έχουμε διευκρινίσει και με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ε, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλετε και αν υπάρχει ζήτημα ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Πάντως αποκλειστικά αφορά μη στρατιωτικές αποστολές. Επίσης, διαπιστώνω με έκπληξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει την κατάσταση κατά τρόπον Απροσδόκητο, γιατί ήμουν ε, και εισηγητής εγώ της Επιτροπής του, ε, ε του προπολογισμού του ορίζοντα 2020 και εκεί πέρα η Επιτροπή ζητούσε εξάπαντος να έχει ε, πράξη συμπράξη και για, τις, ε, για την εκτέλεση του προπολογισμού. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς η Επιτροπή επιδεικνύει μια τέτοια θέση αρχής η οποία άλλωστε δεν μπορεί και να υπάρχει, γιατί είχαμε πει ότι κατά περίπτωση θα βλέπουμε ποια είναι η πιο ευέλικτη και κατάλληλη λύση. Φυσικά πάντα με την επίβλεψη του ελεύθερου προπολογισμού και τη στήριξη των κανόνων. Για τα παραδείγματα τώρα, τα συγκεκριμένα. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ακόμη και ξέρετε ότι κινείστε σε πολύ λεπτό πάγο αν μου λέτε ότι τα πράγματα λειτουργούν ήδη καλά και ότι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι ενδιαφέρον να δούμε και εμείς ε, τι είδου στάση τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Ένα μέρος τουλάχιστον της Επιτροπής. Γιατί και ο ύπατος εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι κομμάτι, ο ύπατος εκπρόσωπος είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορείτε να μου λέτε ότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν το βλέπω αυτό να είναι πολύ συνεπές σαν θέση της Επιτροπής. Και ένα παράδειγμα λοιπόν που μπορεί να διευκρινίσει τα πράγματα στην ε, αποστολή στη Γεωργία που ήταν αποστολή rapid deployment, δηλαδή έπρεπε πολύ γρήγορα να αποσταλούν ε, ομάδες ε, για την περιπολία στα σύνορα. Χρειάστηκε να γίνει διαγωνισμός για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου. και διατυπώθηκε η απέτηση από τις διεθνείς εταιρείε πετρελαϊκών ειδών να εγκαθιδρύσουν ένα δίκτυο προμηθειών, δηλαδή βενζινάδικων το ΣΥΠΗΝ στην περιοχή, για να μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Πρώτα να εγκαθιδρύσουν το δίκτυο και μετά να έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό. Άλλο ένα από τα παράλογα που έχουμε δει και που άλλωστε έχει επικυρώσει και καταγγείλει και το ελεγκτικό συνέδριο. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω την, πρόταση, την ε, ερμηνεία επί της προτάσεως μας. Εμείς παραπέμπουμε στο ελεγκτικό συνέδριο και στα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αποτελεσματικό το σύστημα, καθιονδήποτε τρόπο. Και δεν μπορούμε να απλουστεύουμε σε όρους διαστάσεων, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική, στη δράση, τη μη στρατιωτική, χάνει κάθε αξιοπιστία. Χάνουμε τις φιλοδοξίες και τους στόχους, τους ορθούς στόχους των μη στρατιωτικών αποστολών, διότι δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Είναι γελίο λοιπόν το να λέμε ότι οι διαγωνισμοί, οι διαδικασίες για τις προκηρύξεις και την εκτέλεση του διαγωνισμού κρατάνε περίπου το ίμιση του χρόνου της διάρκειας μιας αποστολής. Είναι παράδεκτο αυτό. Πάντως εμείς από το Κοινοβούλιο και δεν είμαστε διατεθειμένοι τουλάχιστον από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου να ε, το αφήσουμε το θέμα αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε με έμφαση. Το ζήτημα δε των πράξεων και θα απαντήσω ορυτά στο ότι δεν, έχει, δεν είναι ζήτημα συνθήκων, δεν εξαρτάται από τις συνθήκες. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε ένα σύστημα open box ή μια εν επιταγή για δράση. Θέλουμε να μπορούμε να παρακολουθούμε και βέβαια από την σκοπιά της αρχής αρμόδιας για τον έλεγχο του προπολογισμού την εκτέλεση των κονδυλίων. Άρα τα επισήμως προβληθέντα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μένα είναι αβάσιμα. Και καλό τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν με ακρίβεια την πρόταση που έχω διατυπώσει. Νομίζω ότι οι επιφυλάξεις που ετυπώθηκαν έχουν απαντηθεί επαρκώς. Και πάνω απ' όλα, εάν δεν κάνουμε τίποτε αμέσως, γελιοποιούμαστε εμείς και δείχνουμε πόσο άνευ σημασία βρίσκουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Χάνουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας, διότι πολύ σπάνια μπορεί να ξανανοίξει η συζήτηση για δημοσιονομικό κανονισμό. Το επισημαίνω αυτό. Εάν δεν δράσουμε τώρα, για χρόνια, για χρόνια ακόμα θα μείνουμε στο σύστημα όπως ισχύει τώρα και δεν θα μπορούμε να περιμένουμε τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και την υποστήριξη που αναμένω για το μέλλον. Ε, ευχαριστώ κύριε Ο καταλαγός των ομιλητών έχει κλείσει. Τον εξαντλήσαμε. Η προθεσμία λοιπόν είναι 10 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, για την κατάθεση τροπολογιών. Η ψηφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι στις 3 Συνεδριάζουμε εκ νέου. Είναι η δεύτερη συνεδρία μας. Ο κύριος Ζωάν Πολπελομέρος, από τον Άτο θα είναι μαζί μας. Ο Κλοντ Φρανς Αρνό επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ευχαριστώ. Sorry. Α, με τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά μόλις ενημερωθήκαμε ότι στην Νότια Ουκρανία έγινε πυρηνικό ατύχημα. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά ο Πρωθυπουργό ενημέρωσε ότι κάτι συνέβη. Δεν ξέρουμε, δεν έχω άλλες πληροφορίες. τι να πω, ε, δεν θέλω να ανισχύσω τον κόσμο, αλλά είναι μάλλον σημαντικό το θέμα, μπορεί να μα επηρεάζει όλου Εννοείται βεβαίω. Πολύ ωραία, ευχαριστώ που το αναφέρατε λέει Θα ενημερωθούμε πάρα αυτά, εννοείται, και θα ενημερώσω όλου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το αργότερο στην έναρξη της απογευματινή συνεδρίασης. Κύριε Έλερ. Θα ήθελα εκ μέρου ε, του συντονιστή μα κύριου Γκάλερ και τη ε, Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο να θίξω και εγώ το ζήτημα τη παρουσία των βουλευτών που έθιξε η κυρία Λέζινγκ. Έχουμε πολλέ ταυτόχρονε συνεδριάσει. Δεν φταίει η γραμματεία γι' αυτό, γιατί και η Επιτροπή των βιο... της Βιομηχανίας και η Επιτροπή ε, των προϋπολογισμών ε, έχουν ταυτόχρονα συνεδριάσει με πάρα πολύ σημαντικά πακέτα, το πακέτο ε, θέματα όπως το πακέτο Juncker. Εγώ είμαι συντονιστής μάλιστα στην Επιτροπή της ε, Βιομηχανίας. Προφανώς και οι λοιποί συνάδελφοι έχουν ταυτόχρονες συνεδριάσεις, παράλληλες συνεδριάσεις και η απουσία τους δεν σημαίνει αδιαφορία Απλώς θα πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε καλύτερα αν είναι η λύση του να έχουμε παράλληλες συνεδριάσεις με ψηφοφορίες επιτροπών, με πλήρες αρμοδιότητες ταυτόχρονα και να μην μπορεί ο βουλευτής να κάνει τη δουλειά του στην κάθε επιτροπή όπως θέλει. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει να κάνει με την πρόθεση να λάβουμε σοβαρά υπόψη ένα ζήτημα, αλλά με την απλή πρακτική δυνατότητα συμμετοχή των συναδέλφων στην συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ. Θα μας απασχολήσει ασφαλώς στο μέλλον τη Ουκρανία. Θα το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά.